Mes chers collègues, bonjour. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Καλημέρα κύριε Τελίτσκα. Le projet d'ordre du Μπορούμε να εγκρίνουμε το σχέδιο μερίσες διάταξης αν δεν έχετε αντιρρήσεις. Δεν έχετε. Αν δεν έχετε επίση αντιρρήσεις, μπορούμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά της 9η Νοεμβρίου. Δεν έχετε αντιρρήσει, εγκρίνονται και τα πρακτικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, ανακοινώσεις θα κάνω μόλι καταφτάσει ο κύριο Μαρινέσκου για να ψηφίσουμε. Γεια σας κύριε Μπαχ, τι κάνετε. Σήμερα είμαστε φόρμα. Ah oui, hein. Bah, Vim, il partage pas ses biscuits déjà. Καλά, ο Βίμ βάντε κάπου ούτε ένα μπισκότο δεν μου δίνει. Alors, nous allons... Λοιπόν, ας αρχίσουμε τώρα με τις προφορίε και θα επανέλθουμε, κύριε Μαρινέσκου. Για να δούμε λοιπόν, έχουμε απαρτία, κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία, αρχίζει τώρα παρακαλώ. Alors, je vais fermer Πέρας ψηφοφορίας. Ωραία. Έχουμε και απαρτία και απ' όλα για να ψηφίσουμε. Προηγουμένως όμως Επιτρέψτε μου να σας κάνω μια σύντομη ανακοίνωση, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν το συνηθίζουμε, αλλά θα ήθελα επ' να σας πω ότι καταλήξαμε σε πολιτική συμφωνία για τον περίφημο κανονισμό της ΕΑΣΑ μετά από έξι τριμερείς διαλόγους και σημαντικό αριθμό τεχνικών συνεδριάσεων που δεν τις μετράμε πια, ανυπολόγιστος ο αριθμός. Την περασμένη εβδομάδα, όλη τη νύχτα, Τετάρτη προς Πέμπτη, ε, είχαμε σκληρές διαπραγματεύσεις για να καταλήξουμε σε συμφωνία τελικώς στις 6 ώρα και 3 λεπτά ακριβώς το πρωί, μετά από 11 ώρες διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή μας τον κύριο Μαρινέσκου και μπορείτε και να το χειροκροτήσετε. Κύριε Μαρινέσκου, σας ευχαριστώ για το έργο σας, για την αγαστή συνεργασία που είχαμε και βεβαίως όλους τους συμμετέχοντες στο διμερή διάλογο για την εξαιρετική επιμονή τους και εδώ μιλώ και για τους συμβούλους, τους διερμηνείς και ε, ε, τα μέλη της γραμματείας μας και τα μέλη της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας και ο Σβέν που απουσιάζει. Να του τα διαβιβάσετε παρακαλώ. Πάντως η νύχτα ήταν ε, αξιοσημείωτη. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επίτροπο κυρία Μπούλτς, αλλά και τον πρέσβη κύριο Κούλ της Ισδονικής ε, Προεδρίας με το επιτελείο τους. Πραγματικά κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία και ήθελα να το τονίσω εδώ στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ κύριε Μαρινέσκου και πάλι. Ξέρω ότι ήταν και δύσκολο πολλές φορές, αλλά τα καταφέραμε. Θέλετε να πείτε τίποτα. Παρακαλώ, κύριος Μαρινέσκο, ευχαριστώ πολύ για τους συναδέλφους φυσικά. Δύο χρόνια εργαζόμαστε για το θέμα αυτό. Όλο το προσωπικό, οι σύμβολοι των πολιτικών ομάδων και η βοηθή των βουλευτών. Και την γραμματεία φυσικά θέλω να ευχαριστήσω. Παρ' όλα αυτά δεν είναι ώρες αυτές, πέντε ώρες, ξημερώματα για να διαπραγματευόμαστε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Προσωπική άποψη αυτή. Επετεύχθη πολιτική συμφωνία, αλλά δεν τελειώσαμε εδώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έχουμε ακόμα δουλίτσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω τα σημαντικότερα ε, έχουν ε, συμπεριληφθεί από τις προτάσεις του Κοινοβουλίου εννοώ στη συμφωνία. Εκκρεμούν όμως ακόμα κάποια πράγματα και ευχαριστώ πολύ και πάλι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαρινέσκου, λέει η Πρόεδρος. Θα ψηφίσουμε. Αρχής ψηφοφορία. Έκθεση. Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και την κατανάλωση καυσίμου των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Είναι γνωμοδότηση αυτή για την Επιτροπή Περιβάλλοντος και ο συντάκτης της γνωμοδότησης είναι ο κύριος Καπούτο. Παρόν. Εδώ. Ψηφίζουμε λοιπόν. Τροπολογία 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τώρα μαζί θα ψηφίσουμε ένα μπλοκ, ένα σύνολο τροπολογιών 7, 8, 9 4 και 5. 7, 8, 9, 4 και 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται όλες μαζί αυτές. Νορκολογία 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Είναι μικρή διαφορά, στο ελέγξουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά την τροπολογία υπερθών 77 η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 78 υπε. Και contre. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 79 υπέ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία στην τροπολογία 79. Παρακαλώ. Πέρασε. Il est rejeté. Απορρίπτεται. 80. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τσεκ, το, θα το ελέγξουμε λοιπόν. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρασε. Ναι κύριε Βαντεγκάμ, μπορείτε να με πιστεύεστε. Εγκρίθηκε. Όταν λέω εγκρίθηκε, εγκρίθηκε. Λοιπόν, 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 82 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται τροπολογία 83 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται η 10 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται η τροπολογία 11 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Την 12 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Έλεγχο θέλετε, παρακαλώ, αρχίζει η ηλεκτρονική απορρίθμιση της 12. Je ferme le vote. Πέρασε. Εγκρίνεται. Δεύτερη φορά κύριε Παμιβαντεγκάμπ, έτσι. Δεν με εμπιστεύεστε καθόλου. Συνεχίζουμε. 13. Υπέ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογή παριθμών 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 36 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμό 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 44 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. Ας την ελέγξουμε παρακαλώ τη 44. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές απορρίψεται. Η τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, Τελική ψηφοφορία τώρα, ηλεκτρονικά, το σύνολο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε, της αρχής ψηφοφορία. 28 υπέρ, 4 κατά. Συγχαρητήρια κύριε Καπούτο. Εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία γνωματότησή σας. Allez, nous continuons Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Προκλήσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση υποδομών στη συνεργατική οικονομία. Παρουσίαση ε, μιας μελέτης ε, από το θεματικό τμήμα. Ευχαριστώ κύριε Μαρινέσκου. Le département thématique est monsieur το θεματικό τμήμα καλείται να έρθει εδώ στο Προεδρείο, όπως επίσης και ο καθηγητής Ματίας Φίγκερ. Λοιπόν, αυτή τη μελέτη την παρήγγειλε η Επιτροπή μας τον Ιούνιο του 2016 για να δούμε τις επιπτώσεις της συμμετοχικής κινητικότητας, η οποία βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη. Και για να δούμε πώς θα χρηματοδοτηθεί το δίκτυο μεταφορών μας. Η μελέτη ανελήφθη από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, που εδώ εκπροσωπεί ο καθηγητής Ματίας Φίγκερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα σας δώσω το λόγο σε μια πρώτη φάση, κύριε Φίγκερ. και θα μας παρουσιάσετε τα πορίσματα της μελέτης σας και στη συνέχεια το λόγο θα λάβουν τα μέλη της Επιτροπής για να περάσουμε σε διάλογο και μπορούμε να δούμε τόσο τα θέματα της μελέτης και τα συμπεράσματά της, όσο και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε. Κύριε Φίνγκερ, έχετε το λόγο. Για περίπου 20 λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, αλλά θα συνεχίσω στα αγγλικά, γιατί και η έκθεση στα αγγλικά συντάχθηκε και ελπίζω να λειτουργήσει το σύστημα. Ναι. Δέκα λεπτά περίμενα και εγώ τόσο είχα απολογήσει. Οι προκλήσεις της χρηματοδότησης των υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο αυτού που ονομάστηκε συμμετοχική οικονομία, αυτόν τον τίτλο μας δώσανε, μας ανέθεσαν, αλλά ήθελα να κάνω μια σύντομη εισαγωγή για την ψηφο, ψηφιοποίηση, διότι θεωρώ ότι η συμμετοχική οικονομία είναι απλώς επίπτωση της ψηφιοποίησης. Τι προξενεί η ψηφιοποίηση. Έχουμε μια ε, ε, αλυσίδα αξιών η οποία μπορεί να είναι υλική, οτιδήποτε υλικό, όπως ένα κουτί, τρόφιμα ή οτιδήποτε άλλο. Και η ψηφιοποίηση αυτό που κάνει είναι ότι ουσιαστικά δημιουργεί ένα ομοίωμα της πληροφορίας, της υλικής πληροφορίας σε επίπεδο δεδομένων. Αυτό κάνει η ψηφιοποίηση. Αυτό έχει τεράστιες συνέπειες. Πρώτα απ' όλα οι πελάτες, οι καταναλωτές δεν περιμένουν απλώς την ηλική διάσταση, αλλά πιο πολύ δίνουν έμφαση στην άειλη ε, διάσταση. Δηλαδή γίνονται πελάτες όχι ενός βιβλιοπολίου υλικού, υπαρκτού, αλλά του Amazon. Αυτή είναι η πρώτη συνέπεια. Η δεύτερη είναι ότι από, αυτή την ψηφιακή, από αυτό το ψηφιακό επίπεδο μπορεί κανείς να δημιουργήσει νέες επιχειρήσεις, νέα επιχειρησιακά μοντέλα, βάσει των δεδομένων που έχουν ε, ε, δημιουργηθεί με αυτόν τον τρόπο. Η πελάτες μπορούν να αγοράσουν τα δεδομένα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται βάσει αυτών των δεδομένων και να μην υπάρχει καμία υλική υπόσταση. Αυτό έχει τρεις συνέπειες με τη σειρά του ο πελάτης λαμβάνει περισσότερες πληροφορίες και περισσότερη, ε, περισσότερες δυνατότητες, περισσότερη εξουσία στα χέρια του. Έχουν καλύτερη επίβλεψη, επισκόπηση της όλης κατάστασης. Αυτό ισχύει και για την αλυσίδα ε, αξιών, την υλική. Δηλαδή σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη πίεση για την υλική ε, διάσταση. Μπορούν να συγκρίνουν καλύτερα οι πελάτες τα προϊόντα υλικός και αυτό δημιουργεί και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Και κατά τρίτον, η προστιθέμενη αξία μετακινείται πλέον προς το ψηφιακό επίπεδο. Δηλαδή η ψηφιακή αυτή το ψηφιακό επίπεδο ιδιοποιείται ένα μέρο τη αξία και αυτό ήταν και ε, η ουσία του στο, της συλλογιστικής της έκθεσής μας. Εάν η προστιθέμενη αξία βρίσκεται τώρα στο ψηφιακό επίπεδο, το ερώτημα πώς χρηματοδοτούμε τις υποδομές, πώς χρηματοδοτούμε το υλικό επίπεδο, έρχεται ε, σε συνδυασμό με την ψηφιακή διάσταση. Αυτό ήταν το σημείο αφετηρία για τη συλλογιστική μα. Τώρα η έκθεση ίδια. τι μας απασχολεί όταν μιλάμε για συμμετοχική οικονομία. Εδώ έχουμε ένα νέο μοντέλο για την ε, κινητικότητα, αλλά υπάρχει ένα νέο μοντέλο για την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, για όλα τα οποία μπορούν ουσιαστικά να έχουν ένα νομίωμα ψηφιακό. Ε, αυτό που γίνεται σημαντικό είναι οι λεγόμενες ε, διαδικτυακές πλατφόρμες. Τα δεδομένα βρίσκονται σε πλατφόρμες και υπό οικονομικούς όρους μιλάμε για μια αγορά πολύπλευρη του ε, πελάτη που μπορεί να έρθει σε άμεση διάδραση με τον προμηθευτή. Δηλαδή, αν πάρουμε ως παράδειγμα την Uber. Μπορεί κανεί να είναι πελάτης της Uber, αλλά μπορεί να είναι και κάποιο που παρέχει υπηρεσίε βάσει της Uber. Εδώ λοιπόν υπάρχουν ένα σωρό αξίε βάσει της συνεργατική αξίας. Η κατανομή ενός οχήματο, το carpooling, είναι ένα τρόπο, Υπάρχουν όμω κι άλλα. Ε, οι υπηρεσίες κατανέμονται, υπάρχει μοίρασμα των υπηρεσιών. Το να μοιράζεται κανείς το ε, όχημά του είναι κάτι που ε, κάνει ο κάτοχος μοιραζόμενος τις υπηρεσίες με άλλους χρήστες ή ένα ποδήλατο. Έτσι λοιπόν η ε, διαδρομή και το μοίρασμα μιας διαδρομής ε, έχει την εξή διαφορά. Στην ε, περίπτωση της διαδρομής ουσιαστικά παρέχεται και το ε, και στην περίπτωση της, του μοιράσματος διαδρομής Μόνο αν υπάρχει κάποια υπηρεσία που θα πρέπει να δοθεί ε, υπάρχει η κατανομή, το μοίρασμα, ενώ στην περίπτωση του αυτοκινήτου υπάρχει και η υπηρεσία. Ουσιαστικά δηλαδή γίνεται μια διέρεση των δικαιωμάτων. Για όλες αυτές τις πληροφορίες βρήκαμε δεδομένα, τα οποία είναι όλα δευτερογενή. Δεν κάναμε καμία πρωτογενή έρευνα, ουσιαστικά συλλέξαμε πληροφορίες που υπήρχαν ε, ούτως ή άλλως. Μιλάμε για μια έκθεση από την Consult PwC που διαπιστώνει ότι ξεπερνάει περίπου τα 5 δις ευρώ στην Ευρώπη ε, για το 2015 το εισόδημα από την ε, συνεργατική κινητικότητα. Ας προχωρήσουμε λίγο. Το ερώτημα ήταν κατά πόσον το μοίρασμα ενός αμαξιού, η κοινή χρήση ενός αμαξιού μπορεί να υποκαταστήσει τις συμβατικές μορφές μεταφορών. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δηλαδή. Εδώ συγκρίναμε δύο επιχειρησιακά μοντέλα. Ένα είναι το carpooling, το κλασικό μοντέλο είναι το bla car, το οποίο απαντάται στην Γαλλία, την Ισπανία και σε άλλες χώρες και η διάκριση που κάναμε ήταν μεταξύ μεγάλων διαδρομών και αστικών διαδρομών. Για τις μεγάλες διάρκειες διαδρομές είχαμε πολλά άλλα μεν παραδείγματα, θα τα δείτε στην έκθεση, αλλά εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα που συγκρίνει την διαδρομή από το Παρίσι στην Λίλ. Ε, υπάρχουν ανάλογες συγκρίσεις, Βαρκελόνη, Αλικάντε, Παρίσι, Φραγκφούρτη κτλ. Όλα αυτά δείχνουν ότι το carpooling είναι ένα ελκυστικό μοντέλο διότι είναι φτηνό και ως προς τον χρόνο είναι αποτελεσματικό. Όχι τόσο αποτελεσματικό όσο το τρένο, αλλά και πάλι είναι αρκετά γρήγορο. Είναι ένας ελκυστικός τρόπος μεταφοράς και ε, είναι ένας τρόπος να βοηθηθούν όσοι έχουν χαμηλότερο εισόδημα. Αυτό είναι μια συνέπεια από την ε, κοινή χρήση ενός οχήματος για τις ε, μαζικές μεταφορές. Αυτό που βρήκαμε είναι ότι έχει μεγάλες διαστάσεις το φαινόμενο σε κάποιες χώρες, ιδίως στη Γαλλία, και από εκεί κυρίως συλλέξαμε τα δεδομένα. Ε, τα περισσότερα είναι γαλλικά δεδομένα επίσημα, δημόσια. Η κοινή χρήση ενός οχήματος, το carpooling, είναι, έχει κυρίως στόχο να μειώσει τον αριθμό των επιβατών, και, μάλλον έχει ως συνέπεια να μειώνει το αριθμό των επιβατών και το εισόδημα για, τις συμβατικ, συμβατικούς, για τα συμβατικά μέσα συγκοινωνία, τα λεωφορεία και τα τρένα. Οι αριθμοί που έχουμε. 6 ε, δις επιβάτες ένα χιλιόμετρο μεταξύ των οποίων και οι οδηγοί. 12% περίπου των ε, εγχώριων, ε, των εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατών, επιβατών σιδηροδρόμων, ανά χιλιόμετρο. Αυτό έχει οδηγήσει σε μία μείωση των ε, μέσων μαζικής μεταφοράς κατά 6% στη Γαλλία. Λιγότεροι επιβάτες για τους σιδηροδρόμους. Όμως το εισόδημα για τις εταιρείες σιδηροδρόμων, μάλλον η απώλεια εισοδήματος μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη, διότι, αλλά δεν έχουμε αριθμούς από αυτού, ε, μόνο και μόνο γιατί οι προσφορές είναι στις ώρες εχμής, όπου οι, οι τιμές είναι και υψηλότερες για τις εταιρείες σιδηροδρόμων. Αυτή είναι απλώς η αριθμή των επιβατών ένα χιλιόμετρο. Τώρα για το εισόδημα αυτό καθεαυτό, για, τους, ε, για τις εταιρείες ίσως και να είναι μεγαλύτερη απώλεια. Τι συστήνουμε λοιπόν. Το πρώτο, και αυτό ε, διέπει όλη μας την έκθεση, χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες. Τα δεδομένα είναι πολύ αποσπασματικά, ε, είναι από εδώ και από εκεί, δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε ακόμη καλά. Παίρνουμε δεδομένα από παραδείγματα που βρίσκουμε τυχαία. Και αυτό βεβαίω μπορεί να είναι αντικείμενο επίκριση. Δεν είναι τόσο συστηματική η μελέτη μα. Επίση, η δεύτερη σύσταση είναι να υπάρχουν ίσοι κανόνε ε, ανταγωνισμού για όλου. Αυτό που τώρα συμβαίνει δεν ε, γίνεται με ίσους κανόνες, διότι στην ψηφιοποίηση υπάρχει ουσιαστικά ε, η αυτό που ωφελεί τους πρωτεμφανιζόμενους στην αγορά. Αυτοί παίρνουν τα μεγαλύτερα μερίδια της αγοράς, δηλαδή τις ώρες εχμής, εκεί που, κάνα, που είχαν το μεγαλύτερο εισόδημά τους και οι ε, συμβατικές εταιρείες. Και επίσης το θέμα είναι οι πολλαπλές επιδοτήσεις. Δηλαδή κάποιες εταιρείες λειτουργούν με πολλαπλές επιδοτήσεις, διασταυρούμενες επιδοτήσεις οι εταιρείε παίρνουν εισοδήματα από τις πιο επικερδείς γραμμές ε, συγκοινωνίας και από τις πιο επικερδείς στιγμές της ημέρας και καλύπτουν τα σημεία που δεν υπάρχει τόσο μεγάλο κέρδος. Εάν ισχύει το screen skimming δεν θα είναι τόσο εύκολο να υπάρξει αυτή η χρηματοδότηση πλέον. να προσπαθήσω να ολοκληρώσω. Το δεύτερο τμήμα είναι η συνεργατική ε, κινητικότητα στις αστικές συγκοινωνίες. Εδώ τα πράγματα αλλάζουν σημαντικά. Οι αστικές συγκοινωνίες δεν το μελετήσαμε αυτό τόσο πολύ. Παίρνουν πελάτες από τα ταξί, αλλά όχι τόσο πολύ βάσει των πληροφορών που έχουμε από τις ε, μαζικές κοινωνίες, από τα παραδοσιακά μέσα. Διότι στα αστικά κέντρα είναι ακόμα πολύ φθηνότερα τα μέσα μαζικές συγκοινωνίες και υπάρχουν και τα προβλήματα συμφόρησης και ούτω καθεξής. οπότε τα προβλήματα δεν είναι τόσο πολύ των εταιριών. Υπάρχουν άλλα προβλήματα, αλλά όχι για τις εταιρείε τόσο πολύ. Ε, σύσταση λοιπόν για αυτό είναι να προωθήσουμε αυτού του είδους τις υπηρεσίες με νομική βεβαιότητα. Νομική βεβαιότητα για να συμπληρώσουμε τα όσα συμβαίνουν. Αυτό θα μπορούσε να ισχύσει και σε ένα βαθμό και για το carpooling. Διότι σε ώρες ε, μη εχμής, ε, για περιοχέ και σημεία που δεν καλύπτονται καλά από τα μέσα μαζική ε, συγκοινωνία θα μπορούσε να είναι μια συμπληρωματική υπηρεσία. Αλλά το γενικό μήνυμα είναι ότι η συνεργατική κινητικότητα καλό θα ήταν να περιλαμβάνεται σε ένα πλαίσιο ε, δημόσιας πολιτικής και να μην την διαχειρίζονται ε, με τρόπο κατακαιρματισμένο ιδιώτες. Συνολικά λοιπόν, αυτό που βλέπετε στην κουκίδα στη μέση είναι ότι οι υποδομές συγκοινωνιών μακροπρόθεσμα μπορεί να ωφεληθούν από τα εξή. Ε, αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Θα σας το δείξω χωρίς να εξηγήσω. Δυσκολεύομαι λίγο με το κοντρόλ. Ε, α, να το. Να το το διάγραμμα. Ε, Αυτά είναι στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αμερικανικά. Μας δείχνουν ότι ο κόσμος που χρησιμοποιεί τη δυνατότητα της μοίρα, του μοιράσματο διαδρομών, κάποιοι το ονομάζουν ride sourcing ε, services, ε, δηλαδή κάτι σαν το Uber, θα πάρουν αλλού ε, τη δυνατότητα του αυτοκινήτου. Δηλαδή το βασικό μήνυμα είναι ότι κινούμαστε στην κατεύθυνση αντικατάστασης του αυτοκινήτου, του ΙΟΤΑΧΗ και να βγει από το σύστημα ε, του αστικού δικτύου μεταφορών. Δηλαδή ε, το car sharing είναι μόνο μία μορφή ε, που καλύπτει όλες τις προηγούμενες για να φύγουμε από τα αυτοκίνητα. Εάν έχουμε λιγότερα οχήματα θα ωφεληθούν και οι διαδρομές μεγαλύτερης απόστασης και διαρκείας και γενικότερα υποδομέ των, μαζικών συγκοινωνιών. Τώρα, για την ιδιοποίηση τη αξία. Οι διαδικτυακέ πλατφόρμες διαχειρίζονται δεδομένα και αυτό το επίπεδο δεδομένων είναι περίπου 18-30%, σημαίνει μάλλον 18-30% της αξίας των υλικών μέσων. Αυτό παίρνει και το έχουμε δει και στις τηλεπικοινωνίες, στην ενέργεια και αλλού. Εδώ υπάρχει κάποια ιδιοποίηση αξίας και θα έπρεπε κάπως να βεβαιωθούμε ότι τα χρήματα αυτά τα ανακτούμε και επενδύονται στις υποδομές. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρουσίαση και να, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση αμέσως με τους συντονιστές. Ο κύριος Βαντεν Κάμπ, για δύο λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτή είναι η δημοκρατία εδώ στο Κοινοβούλιο. Eh, eh, Θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή Φίνγκερ για τις προσπάθειές του. Τρεις ερωτήσεις έχω. Ερώτηση πρώτη. Όταν άκουσα για πρώτη φορά τον όρο συνεργατική οικονομία, σκέφτηκα μια ρομαντική ιδέα. Ότι θα μοιραστώ το αυτοκίνητό μου με τον Ισμαήλ Ερτούγκ, ας πούμε. Και όταν λείπει θα το μοιράζομαι με τον Ζορς Μέχρι εκεί. Οι πολίτες που γνωρίζονται μεταξύ τους και μοιράζονται με ρομαντικό τρόπο τα αυτοκίνητα και τα ποδήλατά του. Μετά όμω τι είδαμε. Ότι είναι τελείως εμπορευματοποιημένο αυτό. Η Uber βγάζει εκατομμύρια, κάποιοι άλλοι χάσανε μετά εκατομμύρια, ε, τώρα η Uber ίδια έχει χαθεί. Ε, ε, πού είναι η ρομαντική ιδέα λοιπόν της συνεργατικής οικονομίας. και με εσά κυρία Πρόεδρε θα μπορούσα να μοιραστώ το ποδήλατό μου, αλλά έχετε γυναικείο ποδήλατο και δεν μου αρέσει να παίρνω το δικό σας. Άρα, ε, τι γίνεται λοιπόν με τις συγκοινωνίες και την κυκλοφορία στις πόλεις, το carpooling. Είναι εις βάρος των δημοσίων μεταφορών. Εγώ νόμιζα ότι θα ήταν εις βάρος του αυτοκινήτου. Τώρα βλέπουμε τρένα και λεωφορεία που υποφέρουν γιατί ο Κόσμο μοιράζεται τα αυτοκίνητά του. Μα το θέμα δεν ήταν να έχουμε λιγότερα τρένα, λιγότερα αυτοκίνητα στου αυτοκινητοδρόμου. Τώρα πώ το έχουμε καταφέρει έτσι. Και επόμενη ερώτηση, τρίτη. Πρέπει να σας πω ότι είμαι μέγας ε, φίλος και υποστηρικτής των Αμερικανών, αλλά δεν με ενδιαφέρουν τα αμερικανικά στοιχεία, γιατί είναι τελείως διαφορετικά ε, ε, και οι πόλεις τους είναι πολύ διαφορετικές από τις δικές μας. Εμείς έχουμε πιο μικρές πόλεις και μπορεί κανείς να πηγαίνει με τα πόδια και ε, με το ποδήλατο παρά τις τεράστιες εκτάσεις που έχουν στις πόλεις τους οι Αμερικανοί. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει για την ευρωπαϊκή συνεργατική οικονομία. Αυτό με ενδιαφέρει. Σα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σερτούγκ. Στα αγγλικά. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε καθηγητά. Μια ερώτηση έχω. Πάμε λίγο στη διαφάνεια 5. Κάνατε μια σύγκριση ανάμεσα στα διάφορα μέσα μεταφορών και το χρόνο που χρειάζεται κανείς για να διανύσει μια απόσταση. Τρεις ώρες και ένα τέταρτο είπατε για την αεροπορία. Αυτό το παράδειγμα δώσατε. Α, για όχι, όχι άμεση πτήση, γιατί τρεις ώρες και τέταρτο από Παρίσι Λίλη με το αεροπλάνο Α, δεν ήταν η πτήση απευθεία. Ε, αυτό, γιατί δεν το καταλάβαινα. Και κατά τα άλλα έχω και εγώ την αίσθηση ότι μπορεί να είναι για το μέλλον ευκαιρία. Για μικρές αποστάσεις, στην αρχή, στο τέλος μιας διαδρομής. Δεν έχω τίποτα να επικρίνω. Ευχαριστώ. Monsieur Robert Dilleux, c'est à vous la parole. Yes, uh, thank you. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, σας καλή καθήγητη. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με το κεντρικό ερώτημα. Πώς να χρηματοδοτηθούν οι υποδομές ε, στη συνεργατική οικονομία. Έχετε ήδη ε, εξηγήσει ότι η αξία του υλικού στρώματος περνάει σε ένα ψηφιακό στρώμα αλλά στις συστάσεις δεν είδα τι εμείς οι πολιτικοί μπορούμε να κάνουμε για τα επόμενα χρόνια για τη χρηματοδότηση των υποδομών. Πρέπει να φορολογήσουμε περισσότερο. Τι πρέπει να κάνουμε ακριβώς, να αλλάξουμε τη φορολογία που επιβάλλεται στις ε, διαδικτυακές πλατφόρμες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας, αλλά αυτή η μελέτη αφορά τις προκλήσεις της χρηματοδότησης των υποδομών στη συνεργατική οικονομία Εξηγήσατε γιατί πρόκειται για πρόκληση, αλλά δεν ε, μας δώσατε και πολλά στοιχεία για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Πρέπει να επανεπενδύσουμε κάποια ποσά. Και τι θα κάνουμε και με εταιρείε όπως η Μπλαμπλακάρ για παράδειγμα. Εγώ θα ήθελα να ξέρω τι ε, μπορούμε να κάνουμε στις αστικές περιοχές, μιας και το επιχειρηματικό μοντέλο δεν πλήττει τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Και όλες αυτές οι εταιρείε θα ε, θα έχουν ως αποτέλεσμα το πολλαπλασιασμό των επιβατών στα διάφορα αυτοκίνητα. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, πώς θα αντιμετωπίσετε την πρόκληση. Είμαστε ε, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Και είπατε προηγουμένως ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, συγκρίσιμα στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή μήπως ε, αυτά τα στοιχεία πρέπει να στοχοποιηθούν καλύτερα, να στοχευτούν καλύτερα σε εθνικό επίπεδο και σε ό,τι αφορά τους ίσους όρους ανταγωνισμού και τις ώρες εχμής θα δίνατε κίνητρα προκειμένου το μοντέλο συνεργατικής οικονομίας ε, ε, σε ώρες εχμής να ε, προωθηθεί και σε ό,τι αφορά τους ίσους όρους ανταγωνισμού δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα καλά τι εννοούσατε. Θα μπορούσατε να μας δώσετε περιττέρω τη στοιχεία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κράμερ, παρακαλώ. Yeah, Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Τρεις ερωτήσεις έχω τα είπε και ο Κάπ αυτά. Όταν είσαι τρία άτομα σε ένα αυτοκίνητο είναι καλύτερο παρά να έχει τρία αυτοκίνητα με έναν επιβάτη κάθε φορά, τον οδηγό. Αλλά αν το συγκρίνουμε με το ταξί, αυτό είναι δίκαιο ανταγωνισμό. Η Uber ήταν το πρόβλημα γιατί δεν πληρώνουν φόρους. Οι οδηγοί δεν έχουν ε, ε, εκπαίδευση, ε, δεν χρειάζεται να εγγυηθούν τίποτα, γι' αυτό έχουν και φθηνότερε τιμέ στην αεροπλοεία ε, μπορούμε να το κάνουμε με πιο φτηνές προσφορές για άλλους λόγους, γιατί συμπιέζουν το κόστος. Μετά είναι αθέμητος ο ανταγωνισμός αυτός στις μεταφορές. Στο σιδηρόδρομο, ας πούμε, ε, θα πρέπει ε, κάθε σειρμός να πληρώνει για κάθε χιλιόμετρο ε, ένα τέλος. Δηλαδή 100% του σιδηροδρομικού δικτύου πληρώνει τέλη, ενώ 1% μόνο των αυτοκινητοδρόμων έχει διόδια. Προφανώς είναι πιο φθηνό το λεωφορείο. Και το, το 60% των εισπράξεων αποτέλει το επανεπενδύει ο σιδηρόδρομος. Και το τρίτο, είπατε στις πόλεις δεν υπάρχει σχεδόν καμία πιθανότητα. Εκεί που είναι λοιπόν καλές οι δημόσιες συγκοινωνίες δεν έχουν καμία πιθανότητα να επιβιώσουν αυτές οι πλατφόρμες. Συμφωνώ, αλλά εκεί που είναι κακό το δίκτυο έχουν. Γιατί καμιά φορά ε, ο κόσμος δεν έχει τρόπο να κυκλοφορήσει, δεν υπάρχει δικτύωση ε, συγκοινωνίας και ο κόσμος θέλει να κυκλοφορεί. Με αυτό το σύστημα λοιπόν μήπως αφαιρούμε την πίεση από τους πολιτικούς ή να βελτιώσουν τις υποδομές των δημοσίων συγκοινωνιών. Γιατί θα βγουν και θα πούνε ότι δεν συμφέρει, δεν χρειάζεται να κάνουμε αυτή τη πάνη, ε, αφού το έχουν αναλάβει οι συνεργατικοί ε, και οι στοδυνικές, αυτό θα ήταν εις βάρος των δημοσίων ε, μεταφορών. αυτά. Αν συγκρίνω βέβαια το σιδηρόδρομο με το αυτοκίνητο, σας είπα τι γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κραμέρ. Λοιπόν, μπορείτε να απαντήσετε εδώ σε αυτή την πρώτη ομοβροντία ερωτήσεων και μετά οι υπόλοιποι. Ναι, ελπίζω ότι τα κατέγραψα όλα. Κύριε Βάντενκαμπ, ξεκίνησατε με τα ρομαντικά ιδεώδη. Εδώ μιλάμε για εμπόριο και μιλάμε για ένα κόσμο που ζει με το εμπόριο και τις επιχειρήσεις. Ωραίο ακούγεται το συνεργατικό και το μοιράζομαι, αλλά οι πλατφόρμες που είναι από πίσω από, αυτήν την, ε, από αυτό το μοίρασμα έχουν δουλειά. Και δεν είναι απλώς τα δεδομένα, είναι οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται για να βγάλει κανείς κάτι από αυτά τα δεδομένα. Ίσως να είναι μια νέα μορφή επιχείρησης και εμπορικού κέρδους και μια νέα μορφή υποδομής. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Εάν αυτό το επίπεδο των δεδομένων ε, είναι μια νέα υποδομή του αύριο, κάτι που μας οδηγεί σε τελείως διαφορετικό τρόπο νομοθέτησης ε, από το να λέγαμε ότι είναι απλώς εμπορικό. Αυτό δεν το απαντούμε στη δική μας τη μελέτη. Εγώ όμως νομίζω ότι θα χρειαστεί κάπου και ρύθμιση υποδομών στην ε, φάση των δεδομένων. Είναι δική μου, το δικό μου το συμπέρασμα. Λοιπόν, αυτό που μπορεί να μα αποσχολήσει είναι το νέο επίπεδο των δεδομένων και αν θα το ρυθμίσουμε, το διευθετήσουμε ω ε, υποδομή ή ω επιχείρηση εμπόριο. Αυτό είναι νομίζω το θεμελιώδη που πρέπει να αναρωτηθούμε. Μετά, για το ε, επίπεδο της ψηφιοποίησης, ε, το κατά πόσον είναι αυτό εμπορικό στοιχείο. Υπάρχει μια συγκέντρωση, υπάρχουν λιγότεροι φορείς, αλλά στην ψηφιοποίηση υπάρχει αυτό που ονομάζουμε the winner takes it all, αυτός που κερδίζει τα παίρνει όλα στο τέλος. Δηλαδή, αν έχει κανείς κρίσιμη μάζα, έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει ένα μεγάλο μέρος της αγοράς. Αυτό χρειάζεται. Περισσότερη ρύθμιση από την άποψη της ε, εξουσίας στην αγορά εργασία και ούτω καθεξής. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε εταιρεία, αλλά συνήθω οι εταιρείε είναι αμερικανικές γιατί ξεκινάνε πρώτες εξαίρεση είναι η BlaBlaCar που είναι γαλλική, αλλά είναι σπανιότατο. Είναι μια από τις σπάνιες ευρωπαϊκές εταιρείες που έχουν αντίσει σε αυτό το χώρο. Μετά, Δίκιο έχετε. Κάνω αυτήν την ε, βασική διάκριση μεταξύ των μεταφορών μεγάλης απόστασης και των αστικών. Όλη η μελέτη βασίζεται σε αυτήν την διάκριση. Ε, είναι διαφορετικό το τι συμβαίνει στις μακράς απόστασης ε, διαδρομές και στις αστικές, διότι είναι διαφορετικό το κατά πόσο παίρνει κανείς το βασικό κέρδος. Ε, είναι στις αστικές τα ταξί αυτά τα οποία χάνουν κυρίως, αλλά ακόμη και αν πάρουν αυτές οι εταιρείε 18-30% του μεριδίου της αγοράς. Δεν σημαίνει ότι αυτό ισοδυναμεί σε 18-30% του υπάρχοντος ε, των όσων συμβαίνουν μπορεί να είναι καινούργια κίνηση, κυκλοφορία. Μετά είναι το θέμα των σιδηροδρόμων. Και ρωτήσατε πώς συγκρίνονται οι με την Ευρώπη. Δεν συγκρίνονται, διότι είμαστε μια ήπειρος ε, σιδηροδρόμων επί της ουσίας. Οι πόλεις μας είναι διαφορετικές, δεν έχουμε τέτοια αστική εξάπλωση. Και είναι πολλά αυτά που πρέπει να εφαρμόσουμε για να κάνουμε τη σύγκριση. Αλλά δεν έχουμε μόνο αμερικανικά δεδομένα, έχουμε και από ευρωπαϊκές χώρες. Άρα οι βασικές τάσεις είναι ολόιδιες, ίσως να είναι διαφορετικές απλώς οι συνέπειες. Και στις μακράς απόστασεις διαδρομές, δεν θυμάμαι ποιος το ρώτησε και δεν τα θυμάμαι και με τη σειρά, αλλά στις μακράς απόστασεις η βασική σύσταση και νομίζω αυτό θέλετε όλοι ε, να πω ε, συμφωνώ να έχουμε ένα σύνολο συστάσεων, αλλά στι μακράς απόσταση, το βασικό μήνυμα είναι ίσοι κανόνες ανταγωνισμού. Ε, Όμω οι ίσοι κανόνε είναι ήδη πρόβλημα μεταξύ οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών. Δεν ε, οξύνεται απλώς από την ψηφιοποίηση. Υπήρχε ήδη αυτή η διαφορά. Πρέπει λοιπόν να δούμε τη διαλογικότητα, την ε, πολυτροπική μεταφορά για να την πω έτσι, ε, γιατί δεν υπάρχουν ε, ίδια ποσά χρηματοδότηση για όλε τι υποδομέ και η ψηφιοποίηση έρχεται ε, ω ένα διπλέον στοιχείο. Δεν είναι από εκεί η πηγή του προβλήματο. Είναι λοιπόν ο ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφορά ένα θέμα, μεταξύ των διαφόρων μέσων. Η ουσία λοιπόν των συστάσεών μα εδώ είναι να αντιλαμβανόμαστε την κινητικότητα, δηλαδή τι κάνει η ψηφιοποίηση μας αναγκάζει να σκεφτόμαστε με πολλούς τρόπους συνδυασμένα. Σε επίπεδο δεδομένων ε, δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι καινούργοι, είναι οι διάφοροι τρόποι μεταφοράς, τα διάφορα μέσα μεταφοράς που ε, έρχονται και συγκρίνονται μεταξύ τους. Εκεί λοιπόν έρχεται και επιτείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των διαφορών τρόπων μεταφοράς η ψηφιοποίηση. Εσείς ως νομοθέτες πρέπει να έχετε μια πολυτροπική ε, προσέγγιση σε όλα αυτά που να συνδυάζει όλους τους τρόπους. Τώρα πώς χρηματοδοτούμε μότες τι υποδομέ. Εάν τι πλατφόρμε, μάλλον αν οι παίρνουν την αξία. Ε, οι φόροι, η επιβολή φόρων σε εταιρείε που το κάνουν αυτό, μερικέ πληρώνουν ε, όπω η Uber που είναι καταχωρημένη στην Ολλανδία ή BlaBlaCar στη Γαλλία. Αυτό είναι ένα μεγάλο φορολογικό ζήτημα. Και το άλλο είναι η επανεπένδυση σε υποδομές να παίρνουμε τα κέρδη και να τα επενδύουμε. Δηλαδή, έχουμε κάποια παραδείγματα. Στην μελέτη υπάρχει μόνο ένα παράδειγμα από τη Μασαχουσέτη, αλλά ε, μια και έχω ένα παράδειγμα, θα το πω από το Σικάγο, υπάρχει φόρο επί των κερδών τη Uber, 50 λεπτά και προσθέτουν κι άλλα 20, τα οποία πρέπει να επανεπενδυθούν στους, στις δημόσιες μεταφορές, στις δημόσιες συγκοινωνίες. Αυτό είναι λοιπόν κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Η Uber ή η λήφτη ή οποιαδήποτε άλλη να χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτηθούν οι υποδομέ. Και υπό την οπτική γωνία τη προώθηση των ε, μαζικών συγκοινωνιών να ε, φροντίσουμε το φόρο προ όφελο των μαζικών συγκοινωνιών. Είναι εφικτό. Έχουμε μόνο αμερικανικά παραδείγματα, αλλά μπορεί να γίνει και εδώ. Στη ΣΥΠΑ γίνεται σε επίπεδο πόλεων. Δεν γίνεται σε επίπεδο εθνικό. Συνολικά λοιπόν αυτό που χρειαζόμαστε είναι περισσότερα δεδομένα προτού μπορέσετε να νομοθετήσετε, νομίζω χρειάζονται περισσότερε πληροφορίε. Για την ώρα τα πράγματα είναι πολύ φλού για να μπορούμε να καταλήξουμε σε οριστικά συμπεράσματα. Ε, ναι, να ολοκληρώσω λέγοντα κάτι. Έχουμε σχετικά σαφή δεδομένα για την ε, Γαλλία, γιατί υπάρχει μελέτη ήδη από το κράτο. Δεν έχουμε ανάλογη ποιότητα δεδομένων στην Ισπανία, ούτε καν στι άλλε χώρε. Για την Uber έχουμε κυρίω δεδομένα από τη ΣΥΠΑ. Και ε, λέγεται ότι η Uber βοηθάει να ξεφύγουμε από το γιοταχή, όμω και εκεί τα δεδομένα είναι κάπω ασαφή και λέει ότι τελικά καταλήγουμε να έχουμε περισσότερα αυτοκίνητα στου δρόμου. Προτού λοιπόν αποφασίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, πρέπει να έχουμε μια καλύτερη πληροφόρηση. Και συνολικά είναι η, πεποίθη, σαφής μου πεποίθηση ότι η ψηφιοποίηση μπορεί να βοηθήσει αν πάμε στο επόμενο επίπεδο, που δεν είναι η Uber ή η BlaBlaCar. Το επόμενο επίπεδο είναι η κινητικότητα ως υπηρεσία συνολικά. Όλοι οι τρόποι μεταφορών ε, συνδυάζονται. Ε, μπορούμε να δούμε παραδείγματα στην Ευρώπη, στο Γκέτεμπορκ, στο Ελσίνκι, όπου έχουν πάει σε αυτή την κατεύθυνση και αντιμετωπίζουν την κινητικότητα ως μια συνολική υπηρεσία. Αλλά αυτό απαιτεί μια προσέγγιση δημόσια πολιτική στην κινητικότητα, όχι μόνο εμπορική. Οι, εμπορικές, οι εμπορικές εταιρείες, οι ε, επιχειρήσεις, ε, είναι χρήσιμες εάν μπουν κάτω από την ομπρέλα αυτής της δημόσιας πολιτικής και κάποια από τα κέρδη τους χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτήσουμε εάν υπάρχουν ίσοι κανόνε παιχνιδιού για όλου του τρόπου κοινωνία. Και τελευταία παρατήρηση, τα δεδομένα. Οι εταιρείε αυτέ ε, έχουν τεράστιο όγκο δεδομένων και τον παράγουν και αν είναι υποδομή τα δεδομένα πρέπει κανείς να ρυθμίσει την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φίγκερ για τις απαντήσεις σας. Να συνεχίσουμε την συζήτηση ο κύριος Ρικέ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Φίνγκερ για την παρουσίασή σας. Είμαι έκπληκτος γιατί περίμενα κάτι που ε, θα συνδεόταν με το κείμενο και διαβάζω, ε, περίμενα μία απάντηση σχετικά με τις ε, δυσκολίες χρηματοδότησης των υποδομών στη συνεργατική οικονομία. Άκουσα τις ε, πρώτες απαντήσεις που δώσατε. Αναφερθήκατε στις δυνατότητες φορολόγησης και κατανομής των φόρων. Εγώ θα ήθελα παραπάνω στοιχεία όμως, γιατί το πρόβλημα είναι πρώτον. Για ποιες υποδομές μιλάμε, για ποια χρήση των υποδομών και τρίτον, τι τέλει χρήσης των υποδομών. Ε, υπάρχουν οι ψηφιακές υποδομές και υπάρχουν και οι υλικές υποδομές δηλαδή ε, οι, δρόμοι. Και να δούμε πώς θα, ε, θα αντιμετωπίσουμε το φορολογικό θέμα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις ε, δυσκολίες ως προς τη χρηματοδότηση. Δεύτερη παρατήρηση. Κάποιες από τις διαδικτυακές πλατφόρμες ε, αφορούν τα μαζικά μέσα μεταφοράς. Άρα ο διαχωρισμός με το ΙΟΤΑΧΗ δεν είναι τόσο ξεκάθαρος και κυρίως τώρα στο πλαίσιο του μοντέλου μας θα υπάρχει ε, ακόμα περισσότερος ε, συνδυασμός των διαφόρων μέσων μεταφοράς. Και τρίτη ερώτηση, το θέμα της ποιότητας των υπηρεσιών. Δηλαδή, οι διαδικτυακές πλατφόρμες προσφέρουν μια υπηρεσία, υπηρεσίες που δεν υπήρχαν πριν. Δηλαδή, η δυνατότητα να έρθει να με παραλάβει κάποιος ε, στο τάδε μέρος, σε τάδε στιγμή, δεν υπήρχε πριν. Υπάρχει λοιπόν μια προστιθέμενη αξία που προσφέρουν αυτές οι πλατφόρμες. Θεωρείτε αυτό ότι αντιπροσωπεύει ένα κόστος ή πρέπει να το θεωρήσουμε ως ε, ε, ε, απόδοση ως κέρδος. Αυτά είχα να πω νομίζω. Αρκετά ήταν ήδη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρίκε. Η κυρία Ντεμόντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς, ε, διερωτώ με πώς θα χρηματοδοτήσουμε. Και όπως είπατε και εσείς, αναρωτιέμαι κι εγώ εάν είμαστε σε θέση να αντικαταστήσουμε τις δημόσιες μεταφορές με την συνεργατική οικονομία ή τέλος πάντων όπως την ονομάσουμε. Νομίζω η τελος παντων οπως την ονομαζουμε μπορεί να είναι μόνο αρνητική σήμερα. Εφόσον οι δημόσιες μεταφορές δίνουν αναμφισβήτητες εγγύησεις για κάλυψη όλης της επικράτειας και φτάνουν και σε περιοχές ή τέλος πάντων έτσι θα έπρεπε που είναι πλέον απόμακρες. Δίνουν κάποιες εγγύησεις ασφάλειας και μετά θα πρέπει να σκεφτούμε και τα δικαιώματα των επιβατών. Σε ό,τι αφορά την την ε, περίπτωση των ιδιωτών ε, το έχουμε εκφράσει και σε άλλες περιπτώσεις, με άλλες εκθέσεις, λέγοντας και στον τουρισμό λόγου χάρη ότι όταν υπάρχει μια αμοιβόμενη υπηρεσία θα έπρεπε οι κανόνες του παιχνιδιού να είναι ίσοι για όλους. Οι κανόνες του ανταγωνισμού δηλαδή. Για το carpooling εντάξει, αλλά όταν μιλάμε για την ε, κατανομή κέρδους ή εισοδημάτων, περνάμε σε άλλο επίπεδο. Επίση, να κάνω δύο ερωτήσει. Η πρώτη είναι, κατά την άποψή σα, είναι δυνατό να συμπεριλάβουμε τι δημόσιε συγκοινωνίε στην συνεργατική οικονομία χωρί να υπάρξει μείωση τη ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι κρατικοί φορεί. Αυτό θα έπρεπε να σκεφτούμε μελλοντικά εάν υποθέσουμε ότι εντάξει μπορούν να καλύπτονται με συγκεκριμένε υπηρεσίε στι απόμακρε περιοχέ που είναι και πιο αεροκατοικημένε, να συμπεριλαμβάνονται δημόσια δημόσιε συγκοινωνίε στην εργατική οικονομία. Και μετά μιλάμε για δεδομένα, για υποδομέ όχι μόνο ψηφιακέ και για μεταφορέ, αλλά και για υποδομέ προστασία των δεδομένων. Υπάρχει εδώ μια είδηση πριν από 10 μέρε ότι η Uber ε, είχε παραβίαση και υπήρξε πειρατεία σε 57, ε, προφίλ, 57 εκατομμύρια προφίλ χρηστών. Εδώ λοιπόν δεν θα πρέπει να υπάρξει και κάποια εγγύηση ασφάλειας, διότι μέσα από τις πλατφόρμες αυτές ε, έχει κανείς δυνατότητα να μοιραστεί την κινητικότητά του με ένα, αλλά και την πιστοτική του κάρτα και προσωπικά δεδομένα που μπορεί να είναι ευαίσθητα. Πώ μπορούμε λοιπόν να προστατεύσουμε του καταναλωτέ του χρήστε σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντεμόντε. Έχω εγγραφεί και εγώ στον κατάλογο των ομιλητών γιατί έχω πολλές ερωτήσεις. Κύριε Φίγκερ, η πρώτη ερώτηση αφορά τους όρους και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήσατε για την έρευνα. Όταν κοιτάω το έγγραφο, βλέπω τους συντελεστές, τους συντάκτες, των οποίων ε, είστε ε, επικεφαλής, βλέπουμε πρώτο όνομα τον καθηγητή Χουάν Μοντέρο. Δύο επιστολές έλαβα στις 17 Σεπτεμβρίου, τις οποίες έχω εδώ, Σε αυτές τις επιστολές μας λέτε από τον Νοέμβριο του 2014 ο καθηγητής Μοντέρο είναι ε, νομικός σύμβουλος ενός γραφείου που δίνει νομικές συμβουλές στην Uber. Αυτό τι σημαίνει ότι ο κύριος Μοντέρο ήταν ένας από τους ε, δικηγόρους της Uber κατά τη διάρκεια της έρευνας. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε. Πρώτη ερώτηση ήταν αυτή. Ναι. Μπορείτε να μου επιβεβαιώσετε αυτή την απάντηση, την ερώτηση, την ε, πληροφορία. Αυτό ήταν γνωστό. Ο λόγος για τον οποίο επέλεξα τον καθηγητή Μοντέρου με τον οποίο συνεργάζομαι εδώ και χρόνια, έχουμε συντάξει μαζί βιβλία για τις επιπτώσεις ψηφιοποίησης μεταξύ άλλων, επειδή είναι ένας από τους σπάνιους ανθρώπους που γνωρίζει καλά το θέμα και δεν θεωρήσαμε και εγώ προσωπικά θεώρησα ότι ήταν πλονέκτημα να συμμετέχει σε αυτή την έρευνα και όχι πρόβλημα. Άλλωστε, ε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτή την έρευνα και ο κύριος Μοντέρο κυρίως ε, εργάστηκε πάνω στο θέμα των ε, ε, μεγάλων δρομολογίων και όχι στο κομμάτι των αστικών μεταφορών. Άρα αυτό ήταν γνωστό. Άρα μας επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει συσχετισμός ανάμεσα στον κύριο Μοντέρο και την Uber στην έρευνα. Άρα δεν υπάρχει θέμα με αυτή τη συνεργασία. Και θα ήθελα να διαβάσω κάτι, γιατί μέτρησα πόσες φορές ε, εμφανίζεται το όνομα Uber, 131 φορές. 41 φορές εμφανίζεται το όνομα της Blablacar. Θα ήθελα να ε, επανέλθω σε θέμα ουσίας. Χρειαζόμαστε κάποιες διευκρινήσεις. Η έρευνα αυτή αφορά τη συνεργατική οικονομία. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι Uber δεν εντάσσεται στον ορισμό της συνεργατικής οικονομίας. Για ποιο λόγο. Και θα σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Όταν ε, καλώ ένα Uber και ένας επαγγελματίας οδηγός έρχεται να με παραλάβει και με πηγαίνει λίγο παραπέρα, τον πληρώνω για τη συγκεκριμένη διαδρομή. Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκομαι μέσα σε ένα επαγγελματικό όχημα με έναν οδηγό. Άρα δεν βλέπω ποιο είναι ο συσχετισμός ε, με μια υπηρεσία κοινοχρησίας αυτοκινήτων ή carpooling. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό κύριε Φίγκερ και με ανησυχεί γιατί έχω την εντύπωση ότι εσείς εντάσσετε την Uber στην ε, συνεργατική οικονομία παρόλο που δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με κάτι τέτοιο και κάτι άλλο που είπατε προηγουμένως σε ό,τι αφορά τη συνεργατική οικονομία αναφέρατε ότι ο επιβάτης μπορεί και αυτός να γίνει οδηγός. Αυτό όμως δεν ισχύει. Είναι λάθος. Γιατί σε μια τέτοια περίπτωση χρειάζονται άδειες. Και έχω την εντύπωση ότι ε, συγχαίρεται κάποια πράγματα με, ε, και αναφέρεστε στο ε, σύστημα Uber Pop που έχει ανασταλεί στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει πια. Για ποιο λόγο. Έχει ανασταλεί γιατί δεν είναι νόμιμη υπηρεσία. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια σαφή διάκριση ανάμεσα στις λέξεις και τα πράγματα και να χρησιμοποιήσουμε τους σωστούς ορισμούς. Πάντως εγώ στην έρευνά σας αυτό, αυτή τη διάκριση δεν τη βλέπω και είναι αλήθεια ότι η συνεργατική οικονομία ε, πρέπει να ακολουθήσει κάποιους κανόνες, αλλά η Uber δεν ανήκει στη συνεργατική οικονομία. Θα ήθελα να ε, επανέλθουμε στις ερωτήσεις. Έχετε το λόγο για έξι λεπτά. Θα αρχίσω να, να σας ε, απαντήσω. Έχουμε ήδη συζητήσει όλο αυτό το θέμα μέσω ε, ε, επιστολών. Η συνεργατική οικονομία, αυτός ο τίτλος μας επιβλήθηκε, δεν τον επιλέξαμε, είναι ο γενικός τίτλος. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν δύο μοντέλα. Το μοντέλο carpooling, ο συνεπιβατισμός είναι το μοντέλο της εταιρείας BlaBlaCar και σε αυτή την έρευνα μιλάμε για ένα μοντέλο υπηρεσιών, όχι για μια συγκεκριμένη εταιρεία. Μιλάμε για το μοντέλο BlaBlaCar και Uber. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες. Τι σημαίνει το carpooling. Κάποιος οδηγεί, παίρνει ένα αυτοκίνητο και πηγαίνει σε έναν προορισμό και θα το έκανε ούτως ή άλλως και στον δρόμο παραλαμβάνει και άλλους επιβάτες. Κάποιες φορές ε, ε, ε, είχαμε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία 20% των ατόμων που δεν θα κάνανε το συγκεκριμένο δρομολόγιο αν δεν παίρναν κάποιον άλλο μαζί τους. Εγώ έχω την εντύπωση ότι τα διάφορα μοντέλα αυτά σιγά σιγά συνδυάζονται Άρα ε, η διάκριση δεν είναι απαραίτητα βιώσιμη. Ε, ε, μακροπρόθεσμα η Uber θα προσπαθήσει να επιτεθεί στην BlaBlaCar και η BlaBlaCar στην Uber. Ίσως να υπάρχει χώρος για δύο μεγάλες εταιρείες που θα κάνουν τα πάντα. Winner takes all. Και είναι εμπόριο, είναι εταιρεία. Η BlaBlaCar παίρνει 30% ε, προμήθεια. Δεν σημαίνει ότι ο, επειδή ο οδηγό θα έκανε ούτως ή άλλως το δρομολόγιο ε, δεν υπάρχει κέρδος εις βάρος αυτού του οδηγού. Μπορούμε να θέσουμε και ερωτήσεις ε, για το αν τέτοιο μοντέλο είναι πραγματικά κοινωνικού χαρακτήρα. Αλλά θα ήθελα να απαντήσω πρώτα στο ερώτημα του κυρίου Ρικέ. Είπατε ότι δεν ε, δίνουμε σαφή απάντηση στο θέμα της χρηματοδότησης. Δείχνουμε πάντως ότι στην περίπτωση τουλάχιστον των σιδηροδρομικών μεταφορών το πρόβλημα της χρηματοδότησης επιδεινώνεται. Άρα η απάντηση, μια και και σχετικό ερώτημα, η απάντηση είναι ένας καλύτερος συνδυασμός των ιδιωτικών και ε, δημόσιων μέσων μεταφορών. Αυτό μας αναγκάζει να κάνουμε η ψηφιοποίηση και θα μπορούσαμε και όλες να φανταστούμε ένα σενάριο στο οποίο αυτές οι πλατφόρμες έχουν υποχρέωση παροχής υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντας σε κάποιες περιοχές οι οποίες δεν εξυπηρετούνται. Καθήκον μας λοιπόν είναι να συνδυάσουμε όλες αυτές τις υπηρεσίες στα πλαίσια ε, υπηρεσιών κινητικότητας ε, σε αστικό και περιφερειακό επίπεδο, όπως και να είναι, είναι απαραίτητος ένας συνδυασμός και αυτό ακριβώς κάνει το μοντέλο Mobility as a Service. Τα δημόσια μέσα μεταφοράς μπορούν να αντικατασταθούν. Όχι. Όχι, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Πρέπει όμως να συνδυαστούν και σε με άλλα μέσα μεταφοράς και ίσως ε, η ένταξη των πλατφορμών αυτών θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση του κόστου της διαχείρισης ε, συνδρομικών μεταφορών μεταξύ άλλων και δημόσιων μεταφορών γενικώ. Το θέμα αυτό δεν περιορίζεται μόνο στις ε, πλατφόρμες ε, υπηρεσιών ε, κινητικότητα στο θέμα του παρασιτισμού, η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας, όλα αυτά δεν περιορίζονται μόνο στον τομέα των μεταφορών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φίγκερ. Εγώ δεν έλαβα πάντως απάντηση στην ερώτησή μου. Ε, νομίζω ότι δεν καταλάβατε το, πώς λειτουργεί το σύστημα. Με την μπλα υπάρχει ένας διαμοιρασμός των δαπανών, κάτι που δεν ισχύει σε άλλες περιπτώσεις. Και εσείς θεωρείτε ότι τα ταξί εντάσσονται στην συνεργατική οικονομία. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ έχω το έγγραφο σύμφωνα με το οποίο ε, ο κύριος Μοντέρο ήταν ε, ε, δικηγόρος Σούμπερ από το 2014, άρα δεν μπορείτε να μας πείτε το αντίθετο. Υπήρχε μια σχέση ανάμεσα στην Ούμπερ και τον κύριο Μοντέρο. Ναι, βέβαια, υπάρχουν στοιχεία, τα όλα είναι ξεκάθαρα. Θεωρείτε ότι ε, μεροληπτεί αυτή η έρευνα. Όχι. Εγώ νομίζω ότι επικρίνουμε και τα δύο μοντέλο. Εγώ ως πρόεδρος της Επιτροπής ε, θέλω να υπάρχει διαφάνεια, άρα σας έθεσα ε, σχετικά ερωτήματα και επιμένω. εγώ πάντως δεν συμφωνώ με τον ορισμό της συνεργατικής οικονομίας. Για παράδειγμα, η BlaBlaCar εσείς εντάσσετε τα ταξί στην ε, συνεργατική οικονομία. Τα ταξί όμως δεν ε, ανήκουν σε αυτό το μοντέλο, όλοι το ξέρουν. Πώς μπορείτε σε αυτή την έρευνα να βάλετε τα ταξί ε, στην συνεργατική οικονομία. Υπάρχει ένα πρόβλημα ερμηνείας. Όχι, δεν έκανα κάτι τέτοιο. Όχι, τα ταξί δεν ανήκουν στη συνεργατική οικονομία. Οικονομία πάντως είναι και η συνεργατική οικονομία. σε ό,τι αφορά την BlaBlaCar. Κάποιοι οδηγούν, πηγαίνουν κάπου και παίρνουν μαζί τους και άλλους επιβάτες. Προσπαθείτε να διακρίνετε κάτι που εγώ δεν κάνω. Αυτό, αυτή η δυνατότητα υπάρχει γιατί αυτές οι πλατφόρμες ε, δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Είτε ένας οδηγός έκανε ούτως ή άλλως το δρομολόγιο, είτε όχι, μικρή σημασία έχει. Θεωρείτε λοιπόν, κύριε Φίγκερ, ότι υπάρχουν δύο μοντέλα. Το μοντέλο της ε, πλατφόρμας της συνεργατικής οικονομίας και ένα ε, μοντέλο με πλατφόρμες που λειτουργούν με διαφορετικό μοντέλο. Και τέθηκε πολύ ενδιαφέρον ερώτημα σχετικά με τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Πρόκειται για πολύ σημαντικό ερώτημα. Νομίζω ότι και αυτή η διάκριση είναι σημαντικά. Τι ε, ονομάζουμε οικονομική πλατφόρμα και τι ε, ονομάζουμε πλατφόρμα συνεργατικής οικονομίας. Μία είναι απάντηση. Δεν υπάρχει συνεργατική οικονομία με τη ρομαντική πλατφόρμα υπάρχει ε, εμπορική συναλλαγή. Ε, είτε διευκολύνεται η συνεργασία είτε όχι. Δεν υπάρχει συνεργατική οικονομία έξω από κάποια πλατφόρμα ε, που είναι ουσιαστικά μια εταιρεία. Ναι, με αυτό δεν, εγώ δεν συμφωνώ. Μιλάτε για μια πλατφόρμα, ψηφιακή πλατφόρμα που κάνει εμπόριο, αλλά υπάρχουν και ψηφιακές πλατφόρμες που υπάρχουν για να προσφέρουν υπηρεσίες και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένας διαμοιρασμός των δαπανών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φίγκερ που ήρθατε εδώ και παρουσιάσατε την έρευνά σας σχετικά με την συνεργατική οικονομία. Θα τα ξαναπούμε σύντομα και συνεχίζουμε. Allez, nous continuons. Et nous sommes sur... Για να συνεχίσουμε λοιπόν. Θα μας παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του σχεδίου κατεξοδότης πράξης σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσει για σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοείας. Madame Daniela Rosca, où êtes-vous? Η κυρία Ντανιέλα Ρόσκα. Ce n'est pas madame Daniela Rosca qui sera parmi vous et ce sera Δεν είναι το κυρία Daniela Roska. On n'entend pas du tout la commission. Qu'est-ce que vous nous dites? Τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν σας ακούμε. Μιλήστε στο μικρόφωνο, παρακαλώ. Λοιπόν, επαναλαμβάνονται οι εργασίε μα. Μηχανισμός ε, διασύνδεσης το Φεβρουάριο του 2017, το Blending Core, και θα ασχοληθούμε με το, την πρώτη φάση της προκήρυξης του διαγωνισμού, ενώ η δεύτερη εκκρεμή ακόμα δεν έχει λήξει μέχρι τον Απρίλιο του 2018 είναι ανοιχτή. Καλωσορίζω τον κύριο Λιβιέ Σιλά, είστε επικεφαλής του τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών ΜΟΒ που ασχολείται με αυτά τα θέματα. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά περίπου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα ε, ε, του πρώτου αυτού διαγωνισμού blending. Είναι ο πρώτος διαγωνισμός που προκηρύχθηκε με αυτή τη μορφή blending call, λέγεται αυτό. Πάρα πολύ σύντομα, ε, τι είναι αυτό και τι διαφορά έχει από ένα κλασικό διαγωνισμό που προκηρύσουμε. Απλούστατα η χρηματοδότηση, η επιδότηση ε, συνδέεται με όρους. Θα πρέπει να υπάρχει και δάνειο, ε, ισόποσο ε, ή καινοτόμο χρηματοδοτικό μέσο. Δηλαδή, αν επιδοτούμε εμεί κατά 20% θα πρέπει όσοι υποβάλλουν την αίτηση χρηματοδότησης να έχουν 20% δάνειο δότησης ή εναλλακτικής χρηματοδότησης στο στήσιμο του project. Ε, και πέρα από τους κλασικούς διαγωνισμούς που προκυρήσουμε, τώρα θα πρέπει να αξιολογείται και η χρηματοοικονομική τους ε, δυνατότητα, δηλαδή να φέρουν ε, την επιδότηση μαζί με το δάνειο και το χρηματοδοτικό μέσο. Εξού και το blending, δηλαδή συνδυασμός χρηματοδότησης. όλα αυτά λοιπόν φτάνουν ε, σε πιο πρώιμο στάδιο από ότι όταν έρχονται να ζητήσουν μια επιδότηση κλασική. Άρα θα πρέπει να τους αφήσουμε κάποιο χρόνο για να ε, ικανοποιήσουν αυτά τα χρηματοδοτικά αιτήματα. Πώς έχει αλληλουχία. Επιλέγουμε το έργο και στη συνέχεια ε, υπογράφουμε σύμβαση χρηματοδότησης αλλά δεν εκταμιεύουμε τίποτα. Τους αφήνουμε ένα χρόνο να φέρουν την χρηματοοικονομική ρήτρα. Και όταν υπογράψουν το σύνολο της συμφωνίας με το χρηματοδοτικό μέσο τότε και μόνο τότε πληρώνουμε εμεί την αντίστοιχη επιδότηση. Άρα υπάρχει και ένα στοιχείο κινδύνου που αναλαμβάνουμε. Και αν ορισμένοι από αυτούς ε, δεν καταφέρουν να βρουν το ισόποσο ε, δάνειο ας πούμε, εδώ δεν υπάρχει κίνδυνος γιατί δεν τους έχουμε εκταμιεύσει τίποτα και τελικά ε, ακυρώνεται, κυρίστε άγωνη η σύμβασή μας. Άρα, Προκηρύχθηκε λοιπόν για πρώτη φορά αυτή η διαδικασία, ο διαγωνισμός αυτός. Θελήσαμε να καλύψουμε όλες τις προτεραιότητες που συνήθως καλύπτουμε από τους κλασικούς διαγωνισμούς. Ακριβώς για να μην αποκλείσουμε κανένα τομέα. Επειδή δεν είχαμε εμπειρία με τους διαγωνισμούς ε, πολλαπλής χρηματοδότησης, ε, blending και είχαμε το συνηθισμένο ποσοστό συγχρηματοδότησης. Βλέπετε εδώ τις ε, απαντήσεις για τους διαδρόμους της ε, διαδρομές, το RTMS, τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων, καινοτομία και νέες τεχνολογίες και άλλα project που δείχνει διαφάνεια. Το CESAR, το ITS, ε, τις θαλάσσιες λεωφόρους κλπ. Και έχουμε και ένα ενδεικτικό προπολογισμό. Ε, δεν έχουν ακολουθηθεί αυτά τα ποσά ακριβώς, γιατί ήταν δύσκολο να προβλέψει κανείς ποια θα ήταν η απάντηση του κάθε κλάδου ή υποκλάδου, αλλά γενικά καλύπτουμε τις προτεραιότητες πάνω κάτω. Δύο λόγια για τη διαδικασία επιλογής τώρα των projects, των έργων. Voilà. Euh, δεχτήκαμε διπλάσιο αριθμό αιτήσεων. Ο ενδεικτικός ε, προπολογισμός μας αρχικός ήταν ένα δις, 65 αιτήσει λάβαμε για διπλάσιο ποσό. Ε, έγινε αξιολόγηση. Ε, σε δύο χρόνους γίνεται αυτό, όπως και για τους κανονικούς διαγωνισμούς. Από τον εκτελεστικό μας οργανισμό εξωτερική ε, πρώτα αξιολόγηση από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Αυτή η εξωτερική αξιολόγηση επέτρεψε να διατηρήσουμε, να κρατήσουμε 41 ε, προτάσεις με προεπλογισμό 1,7 δις. Σας είπα, ο ενδεικτικός ήταν 1 δις και έχουμε φτάσει σε συστάσεις ε, μετά 39 project Καμιά φορά χρειάστηκε να προσαρμοστεί η διάστασή τους και να ε, αναθεωρηθεί προς τα κάτω το ποσοστό συγχρηματοδότησης, αλλά προσπαθήσαμε όσο γίνεται να στηρίξουμε περισσότερα project με τον προπολογισμό που είχε προγραμματιστεί. Αν δείτε λίγο γιατί ε, έργα πρόκειται, θα διαπιστώσετε ότι ένα από τα πρώτα διδάγματα ε, είναι ότι το blending δεν αποκλεί κανένα είδου ε, προγράμματα και έργα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πιο κλασικές υποδομές όπως ο σιδηρόδρομος ή το ε, ERTMS δεν προσφέρεται να χρηματοδοτηθούν με τέτοιο τρόπο. Το αντίθετο, έχουμε project πολύ ενδιαφέροντα και για το ERTMS και για το κλασικό σιδηρόδρομο, τα παραδοσιακά. Έχουμε και ε, project στα κράτη-μέλη, σε κράτη συνοχή, σε κράτη που δεν είναι στη συνοχή. Από όλα. Έχουμε project 24 κράτη-μέλη συνολικά. Άρα μας δείχνει αυτή η εμπειρία και αποδεικνύει ότι ε, το blending αυτού του είδους η χρηματοδότηση μπορεί να μην προσφέρεται για όλες τις περιπτώσεις, αλλά ε, αποδεικνύεται χρήσιμο και ωφέλιμο για συντριπτική πλειονότητα. Σας είπα ότι είχαμε έναν ενδεικτικό προϋπολογισμό ένα δις. Τώρα θα δείτε από τα ποσά ότι χρειάστηκε να καταβάλουμε κάποια προσπάθεια για το ERTMS. Είχαμε πολλές προτάσεις και ενδιαφέρον εκδηλώθηκε πολύ ψηλότερο από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και εκεί θελήσαμε να κάνουμε μια προσπάθεια, δηλαδή διπλασιάσαμε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό μας. Έχουμε αυτό το περιθώριο ευελιξίας, αυτό δείχνει πόσο ενδιαφέρον έχει συγκεντρώσει αυτό το σύστημα. Ποιοι είναι οι τομείς που υπέβαλαν ε, αιτήσει. Ουσιαστικά και πάλι είναι πολύ μεγάλη αντιστοιχία με τους κλασικούς διαγωνισμούς βλέπαμε την κατανομή στην ε, διευκόλυνση συνδέοντα στην Ευρώπη, ΣΕΦ, το γεγονό ότι υπάρχει διαφορετική χρηματοδότηση δεν σημαίνει μεγάλη διαφορά στι ε, υποψηφιότητε και στα έργα που κατατίθεται. Είναι πάρα πολλά τα σύνδρομακά μαζί με αυτό το ERTMS, μερικά οδικά, μερικά ναυτιλιακά θαλασσία και μερικά ε, της εσωτερικής ε, για την καινοτομία. Θα ήθελα να σας αναφέρω τα έργα, θα τα δείτε σε λεπτομέρειες εσείς, ότι έχουμε πολλά έργα για την ε, ηλεκτροκίνηση. Τρία έργα που αφορούν πολλά κράτη-μέλη, και τα τρία, ε, για να, μπουν, να δημιουργηθούν σημεία ε, φόρτισης αυτοκινήτων και υδρογόνο περνάμε από πιλωτικά προγράμματα ερευνητικά σε ένα βιομηχανικό πρόγραμμα για παραγωγή αυτοκίνηση ε, ε, μετρογόνου ε, και με υγροποιημένο φυσικό αέριο για την εσωτερική ναυσιπλοεία. Αυτά είναι σημαντικά για τα εναλλακτικά καύσιμα και την κινητικότητα με λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα. Ποια είναι τώρα τα επόμενα στάδια. Όπως προβλέπει η διαδικασία, θα υποβάλουμε τα πορίσματα αυτά και τα συμπεράσματα ε, προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού γνωμοδοτήσει η αντίστοιχη Επιτροπή του ΣΕΦ και ελπίζουμε να αρχίσουμε από τον καινούριο χρόνο, την επόμενη φάση. Όπως γνωρίζετε, είχαμε δύο καταληκτικές ημερομηνίες. Μία ήταν τον Ιούλιο αξιολογήσαμε την πρώτη φάση και η δεύτερη δεν έχει εκπνεύσει ακόμα η προθεσμία. Ε, είναι ανοιχτή μέχρι τον Απρίλιο. Παρατάθηκε η προθεσμία και έχει κυρίως στόχο να προσελκύσει περισσότερα έργα, περισσότερες υποψηφιότητες στα εναλλακτικά καύσιμα. Αυτή, η παράταση αυτή ανακοινώθηκε και αποφασίστηκε στα πλαίσια ε, της δέσμης μέτρων για την καθαρή κινητικότητα που εγκρίθηκε πριν από λίγες εβδομάδες έχει σημασία να υπενθυμίσουμε ότι παραμένουν ανοιχτέ όλες οι προτεραιότητες. Έχουμε ένα μικρό περιθώριο λιγμών, 20% ε, του συνόλου του διαγωνισμού, αν έρθουν πολύ καλά έργα για άλλες προτεραιότητες ε, άσχετες με την καινοτομία βεβαίως θα τα μελετήσουμε και αυτά, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα 350 εκατομμύρια που έχουμε επιπλέον να πιάσουν τόπο ε, στα καύσιμα τα εναλλακτικά. Και για να τελειώσω, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε χρηματοδότηση βέβαια, αλλά καλό είναι να έχουμε και καλά προγράμματα, καλά έργα. Γι' αυτό δημιουργήσουμε και ένα σύστημα ε, αρρωγής ε, ένα συμβουλευτικό κόμβο advisory hub για να μπορεί κάποιος να κάνει την ε, αίτησή του να την υποβάλει με σωστό τρόπο. Ε, τα επόμενα αποτελέσματα θα έρθουν το καλοκαίρι του 2018. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίαση και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ο κύριος Ερτούγκ. Όχι, δεν τον θέλετε. Μάλιστα. Ο κύριος Ζήλερ. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Η ιδέα του blending ήταν να υπάρξει ανάμεξη με ιδιωτικό χρήμα, το χρήμα των φορολογουμένων και να μπλεχτεί κάπως με τον ιδιωτών. Αλλά εδώ από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια διάκριση στο τι ονομάζουμε δυτικό επενδυτή. Ε, κατά τη γνώμη μου, ή τουλάχιστον από όσα γνωρίζω εγώ για τι χώρε από όπου προέρχομαι εγώ, τι Βαλτικέ, υπάρχει μικρό ενδιαφέρον από του ιδιώτε επενδυτέ για τι υποδομέ μεταφορών λόγου χάρη για το άμεσο μέλλον. Μερικέ φορέ λοιπόν δεν θέλουν να εμπλακούν. Και θέλετε δική σα την άποψη. Βλέπετε κρατικές εταιρείες να παίζουν αυτό το ρόλο, ε, καλυπτόμενες από το χρήμα των φορολογουμένων. Δηλαδή μέσα κάποιου ομίλου και τελικά να υπάρχει το ίδιο που θα συνέβαινε με τις ε, περιπτώσεις των ιδιωτών. Δηλαδή να βλέπετε δημόσιο χρήμα που μπλέκεται στην ουσία γίνεται blending με δημόσιο χρήμα αντί για ιδιωτών και ο κίνδυνος είναι ο ίδιος για το χρήμα των φορολογουμένων. Αντί να έχουμε πραγματικά την επένδυση από ιδιώτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστούμε και για την παρουσίαση ίσως κάποιες ερωτήσεις αμαθούς αλλά, από την πλευρά ενό αδαούς, αλλά όπως είπε και ο κύριος Ζήλε, το blending που κάνουμε εδώ είναι με εμπορικά μέσα. Αναφέρατε τα έργα υδρογόνου. Εγώ τα θεωρώ ακόμα αρκετά δαπανηρά. Πολύ ακριβά για σήμερα. φαίνεται να έχετε εσείς μάλλον καμιά προσδοκία, καμιά πρόβλεψη ότι οι εμπορικές τράπεζες θα τα δουν και ως οικονομικά βιώσιμα σε ένα τοπίο που ακόμη δεν υπάρχουν υποδομές. Και επίσης θα μπορούσατε να μας πείτε ποια ήταν η συλλογιστική σας όταν είδα την ανάλυση των διαφόρων προθέσεων σας σε διαφόρους τομείς υπήρχε χαμηλός βαθμός επιτυχίας για το βασικό δίκτυο. Νομίζω 7 υπέβαλαν αίτηση για να το υποστηρίξουν. Και θα έλεγα και πάλι ότι για να χρηματοδοτήσουμε τέτοιου είδους blending με εμπορικά ε, μέσα, όλοι είναι υπέρ του βασικού δικτύου, αλλά η ουσία για μένα είναι για τους διαδρόμους να δημιουργήσουμε ένα κόμβο που να είναι κοντά σε μια πόλη, μέσα σε μια πόλη, δηλαδή για σκοπούς εμπορικής χρηματοδότησης, ιδιωτικής χρηματοδότησης να είναι πιο ελκυστικό. Γιατί λοιπόν δεν υπήρχε αρκετό ενδιαφέρον. Υπήρχε ένα στοιχείο πολιτικής που εγκρίνατε ή υιοθετήσατε για να είναι πιο περιβαλλοντική η προσέγγιση και για το ERTMS. Επίσης, ε, επιτυχές, μπορείτε να περιγράψετε τι περιλαμβάνει, διότι όλοι είμαστε πέρα, αλλά είναι και ακριβό. Και δύο τελικές παρατηρήσεις η ερχόμενη τελική ημερομηνία είναι Απρίλιο του 2018. Εσεί είπατε καλοκαίρι. Δεδομένου ότι έχουν έναν αριθμό η ρήτρα χρηματοδότηση για τι συμφωνίε με τι εμπορικέ τράπεζε. Μπορεί τελικά να μα φέρει ω το καλοκαίρι. Θα μπορούμε να δαπανίσουμε. Είναι πολλά τα επιλέξιμα έργα, αλλά το θέμα είναι τη χρονική πίεση θα υπάρξει και επίσης μπορείτε να μας αναλύσετε καλύτερα ένα κάτω μέλο. τέλος πάντων ενδεικτικά, Ποιε χώρε ή από ποιε χώρε υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα για καλύτερα και μεγαλύτερα έργα. Έτσι από περιέργεια, γιατί είμαι Τσέχος και ήθελα να δω πώς θα πάνε οι Τσέχοι. Ευχαριστούμε κύριε Τελίντσκα. Κύριε Κράμερ. ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση επίσης. Και βέβαια η μεικτή χρηματοδότηση, το blending, είναι σήμερα πιο εύκολο από ό,τι πριν από 6-7 χρόνια όταν ήταν πολύ ψηλά τα επιτόκια. Τώρα τα ταμιευτήρια ή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν σου δίνουν ε, το μάλλον αρνητικά επιτόκια έχουν και πληρώνονται για να σου φυλάνε τα λεφτά. Εν πάση περιπτώσει, έχω ερωτήσεις από τη Γερμανία, από τη συγκεκριμένη εμπειρία μου. Παράδειγμα, έχουμε ένα ένα ε, Αμβούργο-Κρακοβία, 900 χιλιόμετρα. Στο σιδηρόδρομο ε, με πολλά λεφτά ευρωπαϊκά στην Πολωνία, εντάξει, αλλά στη Γερμανία μόνο μέχρι το Κότμποτς. Έχουμε 50 χιλιόμετρα κενό που δεν ε, είναι ηλεκτρικό. Άρα έχουμε ε, τρένα, όχι επιβατηγά ε, εμπορεύματα που ε, πηγαίνουν ε, ως δίζελ, όχι ηλεκτροκίνητα και ένα τρένο πολιτιστικό μέχρι το Βρότσλαφ που πάει 350 χιλιόμετρα έτσι. Το κρατήδιο του Βράδεμβουρου ενδιαφέρεται πάρα πολύ να κλείσει αυτό το έλλειμμα που είπαν στην κυβέρνηση, την Ομοσπονδιακή, να χρηματοδοτήσουμε εμεί μελέτη, έρευνα, να γίνει ένα σχεδιασμό. Και βγαίνει ο Υπουργό Μεταφορών τη Γερμανία, Ομοσπονδιακό, και λέει απαγορεύεται απαγορεύεται καν να το προγραμματίσετε ακόμα και αν το πληρώσετε γιατί δεν είναι προτεραιότητά μας. Έχει τέτοια εξουσία ο, ο Γερμανός υπουργό Μεταφορών για να το επιβάλλει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα πρέπει το Βραδεβούργο να πάει στην Κομισιόν. Εκατό εκατομμύρια χρειάζονται και αυτό δεν είναι μόνο διεθνής διάδρομος σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά να κλείσει και ε, το κενό Cottbus Girlies. Αυτό θα είναι καλό και για την τοπική κυκλοφορία. Μας λέτε για την ηλεκτροκίνηση στη Γερμανία. 99% μιλούν γι' αυτό, αλλά εννοούν τα αυτοκίνητα. Και 4 δισεκατομμύρια ευρώ δίνει η κυβέρνηση, η Ομοσπονδιακή, για να υποστηρίξει ε, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και στο στη Σύνοδο Κορυφής για τον Ντίζελ αντί να τιμωρήσει ε, τους ε, μεγάλους ε, εγκληματίες δεν κάνει τίποτα. Εδώ έχουμε ηλεκτροκίνητα ποδήλατα, έχουμε τοπική αυτοδίκηση που δίνει λεφτά για ηλεκτρικά λεωφορεία, έχουμε οδικούς χάρτες για τα ηλεκτροκίνητα ποδήλατα και πάνω από τα Τις μισές ε, εμπορευματικέ ε, μεταφορές της πόλης μπορούμε να τις αντικαταστήσουμε ηλεκτροκίνητα ποδήλατα, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν μέχρι και 250 κιλά το ποδήλατο. Και από το κράτος παίρνουν 0 ευρώ. Ορισμένες πόλεις το χρηματοδοτούν αυτό. Ερώτηση λοιπόν, αν είχαμε πιο έξυπνες περιφέρειες, δήμους και κρατήδια στη Γερμανία για να απευθυνθούν στην Κομισιόν, ακόμα και δεν το θέλει ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Μεταφορών, υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότηση από τα 900 χιλιόμετρα μας λείπουν 50 και 100 εκατομμύρια. Να μας πω, πείτε τι να κάνουν για να τους το διαβιβάσω ή ε, να δώσω τη διεύθυνσή σας να τους τα πείτε εσείς. Θα ήταν μια καταπληκτική ιστορία blending αν θέλουμε να προχωρήσει η ηλεκτροκίνηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κράμερ. Να σας δώσω το λόγο για να προσπαθήσετε να απαντήσετε στο σύνολο των ερωτήσεων. Πολύ σύντομα, μια παρατήρηση και δύο ερωτήσει. Η, πρώτη ερώτηση, η πρώτη ερώτηση, ακούγοντα τι παρεμβάσει των συναδέλφων για το blending, Γιατί με τη χρηματοδότηση, μιλάμε για blending με ιδιωτικό χρήμα. Έτσι πρέπει να καταλάβουμε όμω τη χρηματοδότηση που προέρχεται από δημόσιου φορεί. Διότι καταρχά προέρχεται από δημόσιου, κρατικού φορεί. Μιλάμε για ανάμειξη με το ΕΦΣΥ, το οποίο χρηματοδοτεί Άρα αυτά τα εργαλεία η ΕΤΕ, ε, τα οποία ε, ούτως ή άλλως μιλάνε για ανάμειξη με δημόσιο χρήμα. Ε, αυτό κατάλαβα. Και επίσης το ποσοστό αυτό που αναφέρατε είναι το μέγιστο όριο. Η τρίτη μου ερώτηση είναι και παρατήρηση μαζί. Γιατί κάπως εξεπλάγει ε, στο πνεύμα του blending το θυμάμαι και το έχω αναφέρει σε διάφορες στιγμές εκθέσεις μου προς την Επιτροπή για να υποστηριχθεί, αλλά δεν ήταν προϋπόθεση, ήταν κάτι το υποστηρικτικό. Εδώ είναι λίγο περίεργο αυτό που ακούμε, δηλαδή αν θέλαμε να διευκολύνουμε και να προωθήσουμε κάτι, τώρα ξαφνικά το βάζουμε ως προϋπόθεση είναι αυτό κάτι που συνάδει με το πνεύμα των όσων μέχρι τώρα υπερασπιζόμασταν, που ήθελαν απλώ να υποστηρίξουν και να προωθήσουν κάποια πράγματα. Αλλά όχι να το κάνουν προπόθεση. Ναι, και άλλε ερωτήσεις. Αλλά τώρα έχετε πραγματικά το λόγο για να μπορέσετε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Καταρχάς, τι είναι δημόσιο και τι είναι ιδιωτικό. Τίνουμε να θεωρούμε ότι ένα δάνειο που προέρχεται από την ΕΤΕ, εάν υποκαθιστά χρηματοδότηση από τον προπολογισμό, δεν είναι δημόσιο χρήμα. Διότι η ΕΤΕ αναχρηματοδοτείται από την αγορά κεφαλαίων. Άρα η διαχωριστική γραμμή μεταξύ δημόσιο και ιδιωτικού δεν είναι τόσο αυστηρή. Δεν σκεφτόμαστε το νομικό καθεστώ του φορέα που παρέχει το δάνειο δηλαδή, αλλά τι πηγέ τη χρηματοδότηση ε, αυτή καθ' Ε, υπ' αυτήν την έννοια, ουσιαστικά στο πώς προωθούμε τα 39 από όλα τα έργα, ε, το 1 τρίτο είναι ιδιωτικοί αυτοί που τα προωθούν το άλλο είναι ε, οι δημόσιοι φορείς. Μπορεί να λειτουργούν στην αγορά, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι κρατικά, σημαίνει ότι έχουν και ιδιωτική και δημόσια διαχείριση. Και για τις πηγές χρηματοδότησης βλέπουμε 14 έργα, 14 τη ΕΤΕ, αλλά 20 εμπορικέ τράπεζε να συμμετέχουν στο, πρόγραμμα, στο σύστημα χρηματοδότηση. Δεν είναι πάντοτε δηλαδή βάση δανείου. Πολλέ φορέ υπάρχει μια ανάμειξη με μια εθνική τράπεζα επενδυτική ή εμπορική, αλλά για να απαντήσω πιο συγκεκριμένα στον κύριο Ρικέ, η μεγαλύτερη της Γαλλίας, η οποία είναι η RTMS ε, Trackside ε, Paris Lyon, ε, το μεγαλύτερο μέρο έρχεται από δύο ιδιωτικέ τράπεζε στη χρηματοδότηση. Ούτε από την Κέστε Πάρνη, ούτε από κάποια άλλη εμπορική ή αναπτυξιακή τράπεζα. Έχουμε όλα τα είδη συνδυασμών λοιπόν για το. για το υδρογόνο. Είναι το πρώτο έργο του είδους του, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε. Αλλά μιλάμε για μια περιφέρεια που είναι από πίσω με σκοπού στρατηγική ανάπτυξης, δηλαδή να δημιουργήσει ένα δίκτυο υδρογόνου και σημείων ανατροφοδότησης σε υδρογόνο και ε, σταθμούς ακριβώς ανατροφοδότησης. Μιλάμε για μια εθνική αναπτυξιακή τράπεζα που είναι ο βασικός ε, εταίρος και θα πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί. Για το δίκτυο δίκτυο ε, δεν λάβαμε πολλές αιτήσει και είναι δύσκολο να εντοπίσουμε τη ροή ε, του χρήματος για μια τέτοια δομή κομβική και γι' αυτό δεν ήμασταν τόσο ακριβείς εδώ στα αποτελέσματά μας. Τώρα που θα θέλουμε να κάνουμε στη δεύτερη, μέχρι τη δεύτερη προθεσμία είναι να, ανοίξουμε, να διευρύνουμε λίγο την ερμηνεία του, τι μπορεί να προταθεί για ανάπτυξη στα ενεργειακά καύσιμα ή όχι. Τώρα αυτό που γίνεται είναι αν έχει κανείς ένα έργο εναλλακτικών καυσίμων σε μία προτεραιότητα note θα πρέπει να ε, δούμε κατά πόσο εντάσσεται σε κάποια προτεραιότητα για την ώρα. Ίσως να καταφέρουμε να κάνουμε για τα εναλλακτικά καύσιμα λίγο πιο ελκυστικά για τις πόλεις τα έργα αυτά. Για το ITMS, RTMS, σας ανέφερα τον εξοπλισμό των μεγάλων φορτηγών για το δίκτυο αλλά έχουμε και υλικό από τρεις-τέσσερις εταιρείες που έχει αγοραστεί και κάποιες έχουν ένα πολύ ενδιαφέρον σύστημα στην Ολλανδία όπου δεν το χειρίζεται η ίδια εταιρεία το σύστημα, αλλά η δημόσια διοίκηση που μπορεί να το διαθέσει και σε άλλου εταίρου και αυτό επιτρέπει σε περισσότερε από μία εταιρεία να συμμετέχουν ταυτόχρονα. Να το βρίσκουμε ενδιαφέρον. Για το χρονοδιάγραμμα θα έχουμε δύο φάσει. Τώρα είχαμε τη φάση για την πρώτη υποβολή ε, και θα υπογράψουμε τις συμφωνίες κάπου στην αρχή της ερχόμενης χρονιάς και ως την αρχή του 19 θα έχουμε τη ρήτρα χρηματοδότηση που θα ενεργοποιηθεί και θα υπάρξει, μεταφορά, ε, θα υπάρξει χρηματοδότηση. Μετά η δεύτερη φάση θα κλείσει τον Απρίλιο, τότε είναι η προθεσμία, θα αξιολογηθούν τα έργα κάπου τον, το καλοκαίρι και προς το τέλος του 18 θα αποφασιστούν. Ε, αρχές 19 θα ενεργοποιηθεί η ρήτρα χρηματοδότησης και θα είναι επιλέξιμα μέχρι το τέλος του 2023 αυτά. Για τις ειδικότερε ερωτήσεις, για το έργο της Γερμανίας, δεν θα ήμουν σε θέση να σας απαντήσω τώρα, απευθείας, διότι θα έπρεπε να το μελετήσω λίγο καλύτερα για να σας πω πώς έχει προχωρήσει και πώς ε, μπορούμε να το δούμε από την πλευρά της αρεσιμότητας. Αλλά αν θέλετε να το δούμε διμερώς μετά για να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Για την ηλεκτροκίνητη γραμμή. Μετά για το ποσοστό συγχρηματοδότησης. Εφόσον Δεν ξέραμε τι είδος συγχρηματοδότησης θα χρειαζόταν για αυτό το είδος blending, απλώς ακολουθήσαμε το μοντέλο των κλασικών υποβολών. Δηλαδή 20% είναι το κλασικό ποσοστό συγχρηματοδότησης του κανονισμού ΣΕΦ, αλλά για το ERTMS ήταν 40% για τα σημεία συμφόρησης, για το βασικό δίκτυο ήταν 40 λοιπόν, αλλά επειδή για αυτού του είδους τα έργα έχουμε πολλές αιτήσει, έπρεπε να κάνουμε μια επιλογή. Για τα σημεία συμφόρησης να πιέσουμε, ας πούμε, το, να μειώσουμε το ποσοστό συγχρηματοδότησης. Βλέπουμε λοιπόν μια σειρά από μεγάλα έργα όπου θα προτείνουμε ένα ποσοστό συγχρηματοδότησης 20% αντί για 30%. Πράγμα που θα μας επιτρέψει να χρηματοδοτήσουμε περισσότερα. Και όπως είπα, είναι και ένα τεστ αυτό, είναι μια δοκιμή διότι αν αυτά τα έργα πάνε στα ρήτρα χρηματοδότηση με 20% ε, χρηματοδότηση, αυτό είναι καλό και δείχνει ότι την επόμενη φορά μπορούμε να τα σκεφτούμε διαφορετικά, να έχουμε ένα χαμηλότερο ποσοστό χρηματοδότηση για τέτοιου είδους έργα. Δεν θα είναι δηλαδή αναγκαστικά αυτό πάντα το ποσοστό μα για τη χρηματοδότηση, απλώ ακολουθήσαμε τα όσα προβλέπονταν ε, στον κανονισμό του Connecting Europe Facility. Και τελευταίο, δεν μπορέσαμε να σα στείλουμε την κλασική μα μπροσούρα, το φυλάδιο, διότι τώρα περατώνεται, αλλά πολύ σύντομα θα τη λάβετε στα γραφεία σα. Αν μη τι άλλο, την ηλεκτρονική εκδοχή. Τότε, μάλλον πριν έρθω στο, στη συνεδρία, μόλις, ε, μόλις ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική μορφή, θα δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για όλα τα έργα, για μια σειρά από προγράμματα και ευχαρίστω να σας απαντήσουμε ό,τι ερωτήσεις τυχόν έχετε για οποιοδήποτε από αυτά τα έργα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις σας. Ε, και ολοκληρώσαμε και πριν την ώρα που προβλεπόταν. Αν μπορέσουμε να έχουμε σύντομα το κείμενο, ακόμα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας διαφώτισε για τα θέματα του blending, της μικρής, μικτής χρηματοδότησης, κάτι που ήταν ένα από τα βασικά, θα είναι από τα βασικά σημεία στη σημερινή διατάξη μας τα ερχόμενα χρόνια και για τα επιλέξιμα έργα και θα συνεχίσουμε τώρα την ημερήσια διαταξή μας για την προετοιμασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της πρότασης για την κατεξουσοδότηση πράξη σε σχέση με τις τεχνικές ε, απαιτήσει για σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοείας. Στρέφομαι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήρθατε, κυρία Μποσκέ. Έχετε πέντε λεπτά για να μας δώσετε τις πληροφορίες. Α, τόσο στα γρήγορα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους, αξιότιμοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι υιοθετήσαμε μια νέα προσέγγιση προς τη διακυβέρνηση για να προσεγγίσουμε την επικάλυψη των διαφόρων νομικών πλαισίων σχετικά με τα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοείας. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τις πρώτες πτυχές αυτής της νέας προσέγγισης ε, και την ε, την πρότασή μας για την τροποποίηση της οδηγίας 1629 ε, κάθετος 2016. Να υπενθυμίσω ότι η οδηγία του 16 για τις τεχνικές προδιαγραφές προέβλεπε πιστοποιητικά Φυσικά, ε, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία υπήρχαν διάφορα νομικά πλαίσια για τη διαδικασία και τη λήψη αποφάσεων. Ήταν πολύ δύσκολη η αντιστοιχία ανάμεσα στα πιστοποιητικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ε, ε, Επιτροπής για την Αυσιπλοεία στο Ρήνο. Ε, θεωρήσαμε ότι χρειάζονται ε, ένα πρότυπο για τα 14 ε, για όλα τα σκάφη στο Ρήνο. Εδώ έχουμε ένα σχέδιο ε, πράξεις ε, σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για τα σκάφη εσωτερικής ναυσιοπλοείας ουσιαστικά ακολουθεί την ίδια ε, διαδικασία που ακολουθήθηκε και για την επαγγελματική κατάρτιση για την οποία έγινε ε, παρουσίαση πριν από δύο εβδομάδες και εγκρίθηκε και από το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφοράς. Ε, στο ΣΕΣΝΗ κάνουν αναφορά οι ε, προτάσεις μας και οι τεχνικές ε, προδιαγραφές και τα υφιστάμενα κείμενα. Να επανέλθω λοιπόν στην κατεξουσιοδότηση πράξη. Έχουμε κάνει ήδη το πρώτο βήμα που αφορά τη διαδικασία για το σχετικά με το βάση του άρθρου 280.9 ε, της ε, συνθήκης ε, έχει εγκριθεί τον Ιούλιο. Τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στη σύνταξη της κατεξουσιοδότησης πράξης και καλό θα ήταν να υιοθετηθεί πριν την προθεσμία για την μεταφορά στο Εθνικό Δίκαιο τον Οκτώβριο του 2018. Στην συνεδρίαση με την ομάδα εμπειρογνωμόνων τον Οκτώβριο εξηγήσαμε ότι αυτή η πρόταση τροποποιεί κάποια στοιχεία στα παραρτήματα της ε, οδηγίας και κάποιες μικρές αλλαγές για λόγους ε, συνεκτικότητας και θα ήθελα να εξηγήσω ποιο είναι το περιεχόμενο του προτύπου ε, ES3 στο οποίο αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία. 200 σελίδες ε, αυτό το πρότυπο 500 μάλλον σελίδες και στόχος ε, ήταν η ευθυγράμμιση με τις τεχνικές και κανονιστικές εξελίξεις όπως ο κανονισμός για το τροχαίο ε, υλικό που ε, δεν ήταν έτοιμος όταν δημοσιεύτηκε το πρότυπο του 2015 τα μη οδικά ε, μηχανήματα είναι το αντικείμενο αυτού του ε, προτύπου. Υπάρχουν ε, και οι τιμονιέρες καταγράφησαν κάποια ατυχήματα και σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές θα αποτραπούν κάποια από τα ατυχήματα ε, στις φορτηγίδες. Υπάρχουν και διατάξεις για τα παραδοσιακά σκάφη, για τα συστήματα πυρόσβεσης και για τους ηλεκτρικούς ε, εξοπλισμούς. Στο τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοείας ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις εξελίξεις ε, ε, στο τομέα ΣΕΝ και ΣΕΝΕΛΕΚ, ε, το, την οδηγία για τα εναλλακτικά καύσιμα και ε, βρέθηκαν λύσεις για πολλές από αυτές τις περιπτώσεις που θα είναι υποφελής για το κλάδο της εσωτερικής ναυσιπλοείας και φυσικά η ε, συνάδελφος η Μάγνα που ε, ε, παρακολούθησε όλες τις συζητήσεις και τις διαδικασίες ε, θα είναι εδώ για να με βοηθήσει στο να δώσω απαντήσεις σε κάποια συγκεκριμένα τεχνικά ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρόσκα για αυτές τις εξηγήσει και θα ξεκινήσουμε αμέσως με τον εισηγητή μας Κύριε Μπελέ, καλησπέρα. Σας δίνω το λόγο. Είστε επικεφαλής ε, για την ε, βασική πράξη. Μετά θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές και στη συνέχεια θα ξαναδώσω το λόγο στην Κομισιόν για να απαντήσετε. Κύριε Μπελέ, έχετε το λόγο. Βίβο Μπελέτε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως θα θυμάστε, είχα την τιμή να είμαι εισηγητής για το θέμα αυτό, για τη συγκεκριμένη οδηγία για την εσωτερική ναυσιπλοή και τα τεχνικά πρότυπα. Τριμερής διάλογος, πολύ επιτυχής έλαβε χώρα και ολοκληρώθηκε υπό την προεδρία του τότε Προέδρου κ. Κράμερ της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ για την καλή συνεργασία. Έχω μερικές ερωτήσεις και μερικά σχόλια για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες. Μια τεχνική παρατήρηση πρώτα και δεν θα εκπλήξει αυτό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κάνω εγώ αυτό το σχόλιο. Το Κοινοβούλιο και νωρίτερα είχε εμπλακεί και ήθελε να εμπλακεί όχι στην τελική φάση μόνο, αλλά και στην προπαρασκευαστική φάση. Τώρα είναι περισσότερο θέμα εμπειρογνωμόνων ε, που συνεννοούνται και προετοιμάζουν τις αποφάσεις. Εμείς θέλουμε νωρίτερα να παίρνουμε όλη την πληροφόρηση. Δεν θα εκπλήξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που το λέω εγώ αυτό και το ζητώ. Μερικά τεχνικά ζητήματα για το κεφάλαιο 9, για τις εκπομπές. Ρήπων, καυσαέρια, που είναι η άλλη ειδική ρήπη. Και όπως είπε ήδη η εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προτείνεται προσαρμογή και ευθυγράμμιση στον αντίστοιχο κανονισμό. Συγκεκριμένα για τον αντίκτυπο, στο άρθρο 9.01 ε, αναφέρεται ότι το άρθρο αυτό ορίζει κάποιες γενικές διατάξεις και το πεδίο εφαρμογή. για την έγκριση τύπων ε, κινητήρων και την απαγόρευση ε, ανταλλακτικών κινητήρων. Τι θα πει αυτό ε, σε σχέση ε, με ε, τους κινητήρες οχημάτων που κινούνται εκτός δρόμων. Τι είναι αυτό το πράγμα ακριβώς, τι σημαίνει. Το δεύτερο αφορά τον έλεγχο επιδόσεων των ταχογράφων. Ποια αλλαγή γίνεται τώρα σε σχέση με τα ελάχιστα πρότυπα και τις προαπαιτήσεις. Και αναρωτήθηκα, υπάρχει νομική υποχρέωση να έχει ταχογράφο σε ποταμόπλαιο. Μήπως θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Um, Επόμενο θέμα. Ε, ε, ε, μη επανδρομένα. Από ό,τι κατάλαβα, υπάρχουν κάποιες φορτηγίδες οι οποίες προχωρούν με πρόθεση ή ε, ε, ε, δεν, δεν έχουν ε, πλήρωμα, είναι ρημουλκούμενα ε, κάποια σκάφη, ε, τα τραβάνε κάποια άλλα ή τα, ή τα Υπάρχουν τέτοια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαούνες που τις τραβάνε άλλες μαούνες και δεν έχουν πλήρωμα. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Και μετά η χρήση τέτοιων μη επαδρομένων σκαφών μπορεί να ενέχει επιπλέον κινδύνους ασφαλείας πέραν των όσων ε, έχουμε εξετάσει και αντιμετωπίσει. Αυτές είναι οι σημαντικότερες ερωτήσεις. Τα μη επανδρομένα ποταμόπλια, ε, εκπομπή ρήπων και ε, τα άλλα που σας ανέφερε, τα ταχογράφη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Μπελέτ. κύριε Αρτούγκ, τώρα θέλετε το λόγο. Κύριε Αρτούγκ. Αλλού. Αλλού. Κύριε Αρτούγκ, θέλετε το λόγο. Παρακαλώ. Να vous voulez, d'accord. Alors, ensuite... Δεν θέλει ο κύριος Αρτούγκ. Ο κύριος Κιθ Τέιλορ. Εδώ είμαι και ε, ξύπνιος κιόλας. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας εξήγησε πάρα πολύ γρήγορα το έγγραφο αυτό. Αλλά αυτό που δεν μου εξηγήσετε εμένα τουλάχιστον ήταν για ποιο λόγο ένα εξωτερικό φορέα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι το ΣΕΣΝΗ φαίνεται να έχει τέτοια επιρροή στη λήψη των αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για άλλους ε, τρόπους μέσα μεταφοράς έχουμε την ΕΜΣΑ, την ΕΑΣΑ, την ΕΡΑ που τους έχουμε ορίσει ακριβώς ε, σε συναπόφαση με το Κοινοβούλιο. Από πού και πού τώρα έχουμε το ΣΕΣΝΗ τώρα ε, στην εσωτερική ναυσιπλοεία. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ γρήγορη ερώτησή σας όντως. Άλλος κανείς? Κύριε Λούντγκραντ, θέλετε το λόγο. Όχι, είπα κι εγώ. Ε, λοιπόν, κανένας άλλος. Τρεις ερωτήσεις σημαντικές έχετε. Παρακαλώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ για την πρώτη ερώτηση για τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου για ένα καλύτερα καταρτισμένο προπαρασκευαστικό στάδιο και για μένα είναι καινούργια όλα αυτά διότι έφτασα σε αυτή την υπηρεσία μόλις πριν ε, ε, εγκριθεί η οδηγία αυτή. Ένας χρόνος έχει περάσει μόνος, μόνο ε, ε, η Σέσνη. Νομίζω ότι εργάστηκε ω το δυνατόν ε, ταχύτερα για να προσαρμοστεί με τις νέες ε, απαιτήσεις του 2017 και για να είμαστε έτοιμοι πριν την ε, μεταφορά από τα κράτη-μέλη την μεταφορά της οδηγίας ε, μέχρι το χρόνο τον Οκτώβριο. Προφανώς υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και τώρα ζητήσαμε από την ΣΕΣΝΗ να έχουμε και ένα επεξηγηματικό σημείωμα για τις νέες τεχνικές προδιαγραφές, γιατί Ίσως αυτό το επεξηγηματικό σημείωμα να προετοιμαστεί κατά τη διάρκεια τη χρονιάς και να έχουμε και περισσότερες συναντήσεις εμπορογνωμόνων για να συζητήσουμε το περιεχόμενο, δηλαδή την εξέλιξη των τεχνικών προδιαγραφών. Το όντι είναι πολλή δουλειά και τον Απρίλιο στην Ολομέλεια της ΕΣΝΗ θα υπάρξει συζήτηση για το θέμα της διαφάνειας, για το κατά πόσο να έχουμε όσο περισσότερη διαφάνεια γίνεται. Πρόκειται για μια ενεξελίξη δουλειά. Και απευθείας για το ερώτημα του κυρίου Τέιλορ και μετά θα αφήσω τη Μάγδα Μάρθα να απαντήσει στις τεχνικές ερωτήσεις γιατί δεν υπάρχει τυποποίηση και φορέας τυποποίησης. Νομίζω ότι ο συνομοθέτης αναγνώρισε το γεγονός ότι υπάρχει αρκετή ειδική γνώμη, γνώση στην Επιτροπή του Ρήνου και προσπαθήσαμε ε, ο φορέας τυποποίησης να αφαιθεί ε, στην πρωτοβουλία και υπό την αιγίδα της Επιτροπής του Ρήνου. Εξάλλου, από προηγούμενες οδηγίες, ε, την οδηγία για τα εναλλακτικά κάψιμα στις οποίες συμμετείχα ε, τις διαπραγματεύσεις της, ξέρουμε ότι υπάρχει δυνατότητα να αντλήσουμε και από αλλού με ευρωπαϊκά πρότυπα, πρότυπα και το καθεξής. δεν είναι τελείως αχαρτογράφητο πεδίο όλο αυτό, αλλά στη συγκεκριμένη οδηγία μπορούμε να πούμε ότι θα αντλήσουμε πρότυπα από το ΣΕΣΝΗ και επειδή από το 2015 αυτό ούτως ή άλλως αναφερόταν και ήταν μέρος του παρατήματος 2 της οδηγίας, ευχαριστώ Μάρθα. Ε, ευχαριστώ, καλησπέρα σας. Να ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση για τα μη επανδρομένα σκάφη. Όπως ξέρουμε στις κάτω χώρες υπάρχουν κάποια σχετικά έργα. Πιο πολλοί έχουν να κάνουν με τα θαλασσοπόρα ε, σκάφη, αλλά ξέρουμε και στο Βέλγιο ότι υπάρχει ένα ανάλογο έργο. Μπορεί να έχει τελειώσει μέχρι το 2020 ε, και θα κοιτάξουμε εάν θα υπάρχουν ε, ρημουλκούμενες φορτηγίδες μαούνες οι οποίες ε, δεν θα έχουν πλήρωμα. Θα δούμε γιατί είναι καινούριο. Όσο για τους ταχογράφους και τις σχετικές απαιτήσει δεν είναι υποχρεωτικό στην εσωτερική ναυσιπλοεία. Αν όμως υπάρχουν ταχογράφοι, εν πλώ, θα πρέπει να πληρούν ε, τις προδιαγραφές τις οδηγίες που αναφέρουμε στην 2003 ε, του 2006 όσο για τον κινητό οδικό εξοπλισμό. Γενικός στόχος του κεφαλαίου αυτού ήταν να περιγράψει κάποιους όρους για, τα μη, για τον μη οδικό εξοπλισμό, δηλαδή για τη θέση σε εμπορία των ε, μηχανημάτων και κινητήρων και να δούμε και να δούμε πώς διατίθενται στην αγορά. Επίσης, το θέμα είναι πώς συντηρούνται οι κινητήρες, δηλαδή δεύτερη φάση στην ε, διάρκεια ζωής, στην ύπαρξη της, του κινητήρα από την άποψη της ασφάλειας και της προστασίας. Αυτά από δικής μου πλευράς. Ευχαριστούμε πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που απήντησε στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Να θυμίσω ότι το Κοινοβούλιο παρακολουθεί στενά την προετοιμασία και τη σύνταξη των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Και θυμίζω στην Επιτροπή ότι και εμείς, το Κοινοβούλιο, πρέπει να, να τηρούμαστε διαρκώς ενήμεροι ε, ε, όπως και οι των κρατών μελών. Οπότε θα ε, αναγκαστείτε να μας βλέπετε συστηματικά και ανατακτά χρονικά διαστήματα. Σας ευχαριστώ κύριε Ρόσκα και θα σας πω εις το επανειδήν. Και να συνεχίσω τη συνεδρίαση μου, αλλά και κλεισμένων των θυρών. Να ανακοινώσω ότι θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για να πάυσει και η μετάδοση στο διαδίκτυο και να φύγουν όσοι δεν χρειάζεται να βρίσκονται εδώ από